υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, πρώτη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 52 περνάμε τώρα. 52 σε δύο μέρη. Τώρα ας χρησιμοποιήσουμε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας και ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας. Κλείνει η ψηφοφορία. 21 υπέρ. 21 υπέρ. Ε, κανείς κατά και μία αποχή. Το δεύτερο μέρος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 15 υπέρ, 9 κατά. Άρα εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στο 53. Υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55. Υπέρ κατά αποχές 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ της Ναντιαχής κατά απορρίπτεται 58 υπέρ Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 58. Λίγη. 15 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. 59 υπέρ. Ας ψηφίσουμε. Ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη. 15 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ξεκινήρα ψηφοφορία για το 60. Κατέπεσε το 60. Ωραία. Τότε για, το, για την τροπολογία 61. Ξεκινά ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. 61. Λίγη ψηφοφορία. 18 υπέρ 9 κατά. Εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 ε, ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία λίγη η 16 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Συμβιβαστική τροπολογία Β. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 ξεκινά η ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί. Also, I open the vote. Madame Λοιπόν, ε, ξεκινά ηλεκτρονικά, λίγη ψηφοφορία, 15 υπέρ, 9 κατά. Εγκρίνεται. Ε, 78 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ καταπίπτει, καταπίπτει με συγχωρείτε. Οπότε προχωράμε στην 80. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 80. Λίγη.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 Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 13 υπέρ 15 κατά. 92 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 95 ξεκινά ηλεκτρονικά. Λίγη. Απορρίπτεται 14 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία προφορική 4 ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινά. Λίγη. 13 υπέρ, 14 κατά. Απορρίπτεται. 96. Δεν ψήφισε, είχα ένα πρόβλημα. Τροπολογία προφορική 4 ζητά να επαναληφθεί η ψηφοφορία διότι δεν λειτουργεί στο μηχάνημά του. Οπότε επαναλαμβάνουμε διότι ο κύριος δεν ψήφισε. Προφορική τροπολογία 4. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Πάλι 14 πέρα 14 κατά, άρα απορρίφθηκε. 97 ε, Ξεκινάει ηλεκτρονικά, λίγη, απορρίπτεται. 97 ξεκινά. 97 ξεκινάει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται 18 υπέρ 9 κατά. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, ξεκινώ την ψηφοφορία για την 100 ηλεκτρονικά λίγη απορρίπτεται 13 υπέρ 15 κατά ξεκινά ψηφοφορία για το 101 λίγη επαναλαμβάνεται. 101. Ξεκινά ηλεκτρονικά. Λίγη. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 15 κατά. 102. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 106. Δύο τμήματα ηλεκτρονικά. Ε, ξεκινά πρώτο τμήμα. Λίγη. Εγκρίνεται για το δεύτερο τμήμα τώρα.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 αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 121 ξεκινά η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγοι. 13 υπέρ, 15 κατά, περίφθη. 122. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 123. Λίγη. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 128. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ξεκινά ηλεκτρονικά για την 6 λίγη εγκρίνεται 14 υπέρ 13 κατά ξεκινά ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 7 λίγη εγκρίνεται. Ε, ψηφοφορία ηλεκτρονική για την 8. Λίγη. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της 9. Κατά εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 11. Λίγη. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, 11 κατά. Ποιο είναι υπέρ τη 12. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, ξεκινά ηλεκτρονικά για τη 16. Λίγη. Εγκρίνεται. 17 ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. Απερίφθη. 18. Σε δύο τμήματα ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα. Λίγη. Εγκρίνεται. Ξεκινά ηλεκτρονικά το δεύτερο μέρος. Λίγη.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 μία κατά και δύο αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Μαρία, good work. Mr. Μαρία, καλή δουλειά. Ε, ε, σαν σκιώδης εισηγητής ε, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια Μαρία Μπαντία Κουσέτ και θέλω να πω στους συναδέλφους οι οποίοι Πέβαλαν 134 τροπολογίες ότι υπήρξε πολύ καλή συνεργασία. Τώρα πάμε στην επόμενη. Είναι η πρόθεση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης πρακτικής και μαθητείας. Καταρίνα, Θέλεις το λόγο για λίγο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ηγητές και όσους υπέβαλαν τροπολογίες και θα ήθελα να πω ότι ε, εάν δεν υποστήριξα κάποια πράγματα θέλαμε ένα ε, σύντομο κείμενο το οποίο να είναι όσο γίνεται πιο σαφές. Ευχαριστώ όλους. So, as far, as far as I see, have to vote. Από ό,τι βλέπω θα πρέπει να, ξεκινήσουμε, να ψηφίσουμε με τις κάρτες μου, διότι νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θέματα αμφιλεγόμενα. Εάν υπάρχει κάποια τροποποίηση στον κατάλογο των, ε, ψηφοφοριών, να το πείτε στους ε, συναδέρφους. Όταν φτάσουμε δηλαδή στις μεμονωμένες τροπολογίες. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 2. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, αρχή της ψηφοφορίας για την τρία ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Ποιος είναι υπέρ της 4. Κατά. Εγκρίνεται. 5. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχή της ψηφοφορίας για την 6. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ποιος είναι υπέρ της 7. Κατά. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της 8. Κατά. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται. Ποιος είναι υπέρ της 10. Κατά. Απορρίπτεται. Ποιος είναι υπέρ της 12. Κατά. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 15. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχή της ψηφοφορίας για την 16. Όλοι είναι υπέρ νομίζω. 16. Λήξη της ψηφοφορίας. Ναι, ευχαριστώ. Αρχή της ψηφοφορίας για την 17. Λήξη της ψηφοφορίας. Τέλεια. Ε, εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της 18. Κατά. Απορρίπτεται. Αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 19. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ποιο Ποιος είναι υπέρ της 22. Ε, κατά. Κανένας εσάς εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αρχή της ψηφοφορίας για την 24. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται αρχή της... Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Ποιος είναι υπέρ της 25. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, 28, συγγνώμη, 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 29. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ποιος είναι υπέρ της 30. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35 αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της 37. Κατά. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της 38. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45. Αρχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αρχή της ψηφοφορίας για την 47. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, αρχή της ε, ψηφοφορίας για την 48, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 49, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Υπέρ της 50, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 51. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 52. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της 53. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία την 55. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ποιος είναι υπέρ της 57. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπέρ της 58. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπέρ της 59. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αρχή της ψηφοφορίας για την 60. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ποιο είναι υπέρ τη 61. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Ε, τελική ψηφοφορία. Αρχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Νερεδαλόα, ήταν η πρώτη σας έκθεση. Ο κύριος Φίσας. Just to congratulate. Να συγχαρώ την Κατερίνα Νεβετάλοβα για την καλή της ε, έκθεση, την καλή συνεργασία και για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. So, wir kommen jetzt zu Punkt 9 der Tagesordnung. Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Ο συνάδελφος Λίγκεκαρτ Äh, ο συνάδελφος Λούκεγκάρτ θα παρουσιάσει την ε, έκθεσή του ε, με τίτλο σχετικά με τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα ενημέρωση δημιουργία μια δημόσια σφαίρα στην Ευρώπη. Είναι έκθεση πρωτοβουλία και τη συζητήσαμε σύντομα το Φεβρουάριο. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριο Λεγκάρτ στην ε, συζήτηση προβλέπει την παρουσίαση ενός εξωτερικού πυρογνώμονα για ένα ημερολόγιο νέων της Ευρώπης το οποίο αποτελεί παράδειγμα του πώς μπορούν τα νέα μέσα ενημέρωσης να βοηθήσουν τους νέους να ε, επικοινωνούν μεταξύ τους. Θα έχουμε λοιπόν τώρα χρόνο για μία σύντομη παρουσίαση. Έχουμε μία ώρα συνολικά. Ε, νομίζω θα την ε, εκμεταλλευτούμε. Ε, προτείνω πρώτα να ξεκινήσει ο κύριος Λέκεγκαρτ και όποιος άλλος ενδιαφέρεται να υποβάλει τροπολογία, ε, τροπολογίες να ξέρει ότι 4 Μαΐου στις 12 η ώρα είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Και θα, συζητήσουμε, και θα, ψηφίσουμε ε, εδώ στην Επιτροπή μας σε 1η και 2η Ιουνίου. Κύριε Λίγα Κάρντ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ε, χαίρομαι που είσαστε τόσοι παρόντες εδώ σήμερα. Χαίρομαι για όλους όσους έδειξαν ενδιαφέρον για την έκθεσή μου. Είναι θέμα σημαντικό όχι μόνο για τα μέλη της Επιτροπής μας, αλλά και για το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ε, κατά τη γνώμη μου διακυβεύονται πολλά. Η μελλοντική επιτυχία του ε, εγχειρήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όλα αυτά εξαρτώνται όχι μόνο από το δυναμικό, αλλά και τη δυνατότητα επικοινωνίας και τη δυνατότητα να συζητώνται τα υπέρ και τα κατά σε ένα διαφανές πλαίσιο. Πολλά έχουν υποθεί κατά τη διάρκεια των ετών για το πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο πολύ εμπειρογνώμονε στην επικοινωνία. Βασικά όμως το πρόβλημα παραμένει. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε νέα κατανόηση της πρόκλησης αυτής και χρειαζόμαστε δράση. Η έκθεσή μου προσπαθεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή και να αντιμετωπίσει τα δύο βασικά ερωτήματα. Ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. έχω υποφεληθεί από την ε, ε, αναλυτική γνώση της Κομισιόν ε, στο θέμα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτρόπο και την ομάδα της. Οι συναντήσεις μας ήταν επικοδομητικές και μας ενέπνευσαν πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εσκιώδης ηγητές που είχα τη δυνατότητα να συναντήσω μέχρι τώρα. Ήταν πολύ χρήσιμη η συμβολή σας και οι προτάσεις σας και ελπίζω να συναντηθώ με όλους σας πριν την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών για να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς ε, για το θέμα αυτό. Θα ε, αναφερθώ τώρα στην έκθεση και αυτό το θέμα θα το συζητήσω στα τανέζικα. Όπως είπαμε, η βάση για την έκθεση αυτή είναι σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ε, στον... η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα από, τον... από την εθνική σφαίρα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το πρώτο που θα ήθελα να πω όσον αφορά την επικοινωνία ε, είναι ότι στην έκθεσή μου κάνω διάκριση ανάμεσα στην την πληροφόρηση ε, από την οποία έχουμε πάρα πολύ, μεταξύ άλλων και στα συστήματα εδώ στις ε, Βρυξέλλες, και την επικοινωνία που είναι διμερής, δεν είναι μονοπλευρή όπως είναι η πληροφόρηση. Και κατά τη γνώμη μου λείπει η επικοινωνία. Η επικοινωνία έχει τρεις αποστολείς, τρία κανάλια. Έχουμε τους πολιτικούς, ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα τρία αυτά κανάλια θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία ε, μιας δημόσιας ε, ευρωπαϊκής σφαίρας όπου θα συζητιέται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη δημόσια αυτή σφαίρα ε, θα πρέπει να πραγματοποιείται η επικοινωνία αυτή και διαπιστώνω στην έκθεσή μου ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν μια εθνική δημόσια σφαίρα ε, που δεν περιλαμβάνει στο βαθμό που θα ήθελα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή λειτουργεί καλά. Αλλά μας λείπει μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την απουσία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και επίσης την απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εθνικές δημόσιες σφαίρες. Πώς μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και πώς μπορούμε να κάνουμε την συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι καθημερινό στις ε, εθνικές δημόσιες σφαίρες. Ε, τους μήνες που ασχολούμαι με αυτό, τρία πράγματα ε, ήταν σαφή για μένα. Πρώτον, δεν υπάρχει κάποια εύκολη λύση διότι εάν υπήρχε θα την είχαμε βρει ε, μέσα στα 50 χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Χρειάζεται ένα μπουκέτο, χρειάζεται ένα, μια γκάμα ε, διαφόρων λύσεων. Το άλλο που συνειδητοποίησα είναι ότι λείπει πολιτική ηγεσία. Ε, λείπει πρωτοβουλία από την κορυφή για το θέμα αυτό και γι' αυτό έχουμε την κατάσταση που διαπιστώνουμε όπου η κορυφαίοι πολιτικοί κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα πράγματα πάνε στραβά, ενώ όταν τα πράγματα ε, πάνε καλά καρπώνονται οι ίδιοι τους επένους. Ε, χρειάζεται λοιπόν πολιτική ευθύνη. Το τρίτο πράγμα που συνειδητοποίησα κατά τη διάρκεια τη διαδικασία αυτή είναι ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια προσέγγιση bottom-up, από κάτω προ τα πάνω. Ε, θα πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε από του πολίτε και να εργαστούμε προ τα πάνω. Έτσι είναι τα πράγματα και αυτό βέβαια περιπλέκει τα πράγματα. Αν κοιτάξουμε την ίδια την ε, έκθεση, ε, προσπάθησα να την χωρίσω σε έξι μέρη. Έχουμε το πολιτικό τομέα. Εδώ είναι περιορισμένο το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως κοινοβούλιο ε, όσον αφορά την πολιτική δομή. Ωστόσο είναι σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός και να πιέσουμε το εθνικό πολιτικό επίπεδο και κοινοβουλευτικό επίπεδο να στο πρόβλημα. Δύο, σημαντικοί δύο σημαντικές παράμετροι υπάρχουν. Χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή από τους πολίτες. Η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να σημαίνει ότι οι πολίτες θα συμμετέχουν πολύ περισσότερο στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί κάθε πέντε χρόνια να περιμένουμε στις ε, εκλογές ε, για το Ευρωκοινοβούλιο ξαφνικά ο κόσμος να ξυπνάει και ε, κατά τα άλλα απλά να ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν κάποιος, έχει καταχραστεί, όταν κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταχραστεί ε, πόρους του Ταμείου. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να γίνει πολιτικό θέμα. Ε, θα πρέπει θα πρέπει οι πολίτε να συμμετέχουν σε, στην ε, λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ε, σε εθνικό επίπεδο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σπρώξουν για να ε, λαμβάνονται αποφάσεις ε, όπου οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων αυτών. Ε, παράδειγμα, η εκλογή του νέου Προέδρου ε, για, του Συμβουλίου και της Υπουργού Εξωτερικών. Εάν αυτοί είχαν εκλεγεί ε, ε απευθείας, ε, τότε θα υπήρχε δημόσιος ευρωπαϊκός χώρος όπου θα, συ, συζητιόταν το θέμα αυτό. Αλλά δεν έγινε έτσι το θέμα. ρυθμίστηκε και κλεισμένον των θυρών. Και νομίζω ότι έτσι ε, ο κόσμο δεν συμμετέχει σε αυτά που συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση θέλουμε περισσότερη συμμετοχή από τα εθνικά κοινοβούλια. Η συνθήκη τη Λισαβόνα ευτυχώ ε, αποτελεί ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για την επικουρικότητα και για τι πρωτοβουλίε των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο επικροτούμε και το κάνω αυτό σε κάποιε παραγράφου. Το δεύτερο μου θέμα είναι τα μέσα ενημέρωσης είναι γεγονός ότι λείπει κάλυψη. Η σοβαρή πλευρά του τύπου στην Ευρώπη ασχολείται σε ικανοποιητικό βαθμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως στην τηλεόραση υπάρχουν προβλήματα. Και δεν μιλάω καν για το εμπορικό κομμάτι, διότι γι' αυτό δεν έχουμε απόψεις. Μπορούμε να έχουμε άποψη, αλλά δεν μπορούμε να, ε, να παρέμβουμε. Αλλά τα ε, τηλεοπτικά κανάλια ε, σε, στις περισσότερες χώρες ε, δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα τα οποία θα αναφέρω, αλλά γενικά υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Και βέβαια εμείς ως πολιτικοί δεν θα πρέπει να παρέμβουμε στην στην συντακτική δουλειά των δημοσιογράφων και ως φιλελεύθερος δεν θα μπορούσα ε, να ε, παρέμβω και στην αγορά. Αντιστρόφως όμως θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε υποχρέωση σε πολιτικό επίπεδο να σκεφτούμε δημιουργικά και να βοηθήσουμε να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και την ε, μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε πολλές συζητήσεις. Η πρόταση 17, η ιδέα δηλαδή να δημιουργηθεί ανεξάρτητη ομάδα δημοσιογράφων ε, η οποία ε, θα καθοδηγείται από, την Ευρωπαϊκή, από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και που θα δημιουργήσει νέα ατμόσφαιρα όσον αφορά την ειδησογραφική κάλυψη θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες πλατφόρμες και κανάλια. Αυτό θα είναι βέβαια πείραμα, θα είναι νέο και ναι θα είναι διασυνοριακό. Δεν αποτελεί προσπάθεια να ε, ε, καταστήσουμε ανέργους τους δημοσιογράφους των Βρυξελών. Όχι, του αντίον. Η ιδέα μας είναι με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουμε περισσότερη προσοχή, περισσότερες ε, καλές, περισσότερα καλά ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες και έτσι να έχουμε περισσότερη προσοχή, κάτι που θα πιέσει, πιστεύω, περισσότερο τις, ε, ε, τους συντάκτες των εφημερίδων να ασχοληθούν περισσότερο με τα, θέμα αυτά, με τα θέματα αυτά. Ούτως ή άλλως υπάρχει σημαντική πίεση από τις ε, πατρίδες των δημοσιογράφων επειδή πρέπει να γίνουν περικοπές. Εμείς μπορούμε όμως να πετύχουμε περισσότερη, περισσότερη προσοχή, περισσότερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα τους βοηθήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό το πείραμα αυτό και ε, για να δούμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσει όσον αφορά την ορατότητα, την ε, διαφάνεια και την ε, σωστή ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήθελα να πω για την παράγραφο 17 και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, Έχω κάποιες προτάσεις για τα τηλεοπτικά κανάλια και τις δημόσιες υπηρεσίες. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχω στόχο να παρέμβω στις επιλογές των ε, ιδιωτικών ε, ε, των καναλιών και εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν θα μπορούσα καν να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Είναι σαφές όμως ότι με το να τονίσουμε, να πιέσουμε απέναντι στις, στα τηλεοπτικά κανάλια αυτά, να επιστήσουμε την προσοχή τους στο πρόβλημα, έτσι δημιουργούμε κάποια πολιτική πίεση. Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα σχετικά με το πώς ε, τα δημόσια κανάλια ε, χειρίζονται το θέμα και γι' αυτό είμαι διατεθειμένος ε, να συμμετάσχω στη συζήτηση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε το θέμα αυτό για να καλύπτονται οι απόψεις όλων, αλλά πιστεύω πράγματι ότι πρέπει να γίνει κάτι στον τομέα αυτόν. Όσον αφορά το σημείο δεν θυμάμαι ποιο, ε, ε, τι, αριθμό έχει. Πάντως εκεί που μιλάμε για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Ε, εξετάζω τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ. Και θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Την ιδέα η Κομισιόν να οικοδομήσει πάνω στην επιτυχία των Scoreboards στην εσωτερική αγορά. Διαπιστώνω ότι ήταν μια από τις επιτυχείς ιστορίες όσον αφορά την ε, ορατότητα και τη διαφάνεια. Και έτσι λοιπόν ε, έχουμε ασκήσει θετική πίεση στα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι η ίδια ε, αρχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί απέναντι στα δημόσια κανάλια για να εξετάσουμε σε τι βαθμό καλύπτουν θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μπόρεσα να δω τα νούμερα που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα στοιχεία αυτά. Καταθλιπτικά αναγνώσματα είναι τα στοιχεία αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα δημιουργώντας ένα scoreboard, έναν πίνακα αποτελεσμάτων. Επίσης, γνωρίζω και θα ήθελα να ε, υπερασπιστώ την πρόσληψη εξωτερικών δημοσιογράφων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε έναν μηχανισμό με με τους συμμετέρους. Ε, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους απ' έξω για να έχουμε νέο αίμα σε μια τέτοια ομάδα. Υπάρχει και το σημείο όπου αναφερόμαστε στο τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις δράσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτών. Ε, γίνονται συμφωνίες για περιφερειακά ραδιοφωνικά κανάλια. Το πρόγραμμα αυτό μόλις έχει ξεκινήσει και ε, το φθινόπωρο θα ξεκινήσει μια συμφωνία για ε, περιφερειακή τηλεόραση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και έτσι μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση bottom-up από κάτω προς τα πάνω και να εξετάσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν με τα εθνικά δίκτυα και έτσι να τα παρακάμψουμε. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να γίνει σημαντική προσπάθεια στον τομέα αυτό. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι για να διατηρηθεί αυτό, επειδή είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία των συντακτικών ομάδων που θα ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Αυτό πρέπει να το ξανατονίσω, διότι αλλιώ δεν θα έχει καμία αξιοπιστία ένα τέτοιο, πρόγραμμα. Πάντω το στηρίζω με όλη μου την καρδιά και <clears throat> ελπίζω ότι θα μπορέσει αυτό να συνδεθεί με την πρωτοβουλία που αφορά την Task Force, την ομάδα κρούση των δημοσιογράφων. Πρώτο θέμα, η νέα τεχνολογία στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα, διότι εδώ μπορούμε να ελπίζουμε σε σημαντικές ε, βελτιώσεις. Τα πράγματα με τα οποία έχω ασχοληθεί μέχρι στιγμή στην ε, έκθεση είναι πράγματα που, ε, ε, τα οποία μπορούμε να επηρεάσουμε μόνο ε, σε βαθμό, διότι, ε, μόνο, μέχρι, μόνο σε κάποιο βαθμό, διότι αυτά είναι πράγματα που ήδη υπάρχουν και δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην αγορά. Αλλά όσον αφορά τα κοινωνικά μέσα ενημέρωση, εδώ μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλά. Ειδικά στο Κοινοβούλιο κάνουμε πολλά πράγματα και η Κομισιόν θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Σημαντικό είναι ότι Ε, τα κοινωνικά αυτά μέσα ενημέρωσης, το Facebook, το Twitter και άλλα. Σημαντικό είναι ότι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά ε, η προσέγγιση bottom από κάτω προς τα πάνω φαίνεται να είναι δημιουργημένη ειδικά για τα μέσα αυτά. Μπορούν λοιπόν να γίνουν πολλά. Θα ήθελα να υπερασπιστώ και εδώ τις κοινοπραξίες σε δημοσίου ε, ιδιωτικού τομέα. Όταν κοιτάμε τα πλαίσια αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική γνώση, σημαντική τεχνογνωσία σχετικά με την επικοινωνία στα πλαίσια των κοινωνικών μέσων ενημέρωση και του διαδικτύου το, και το πώς γίνονται κοινοπραξίες ε, στον τομέα αυτών. Και γι' αυτό σήμερα ε, ήθελα να σας παρουσιάσω ένα παράδειγμα για να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, τι ακριβώς συμβαίνει και επίτηδες επέλεξα ένα παράδειγμα το οποίο απευθύνεται στους νέους, διότι αυτοί αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση. Ε, δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με την ομάδα ηλικίας 15 με 25 ετών, το οποίο σημαίνει ότι από πολιτικής πλευράς είναι πολύ χρήσιμο να ε, ε, λάβουμε εμπειρίες απ' έξω. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο σε έναν εκπρόσωπο ενός προγράμματος με το οποίο είχα κάποιες εμπειρίες για να σας δείξω τι ακριβώς γίνεται στον τομέα αυτόν. Ε, παραγωγός ε, ταινιών που λέγεται Copenhagen Bombay, ε, Bombay, ε, έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα όπου συμμετέχουν οι νέοι, είναι συμπαραγωγή οι νέοι. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία και θα έπρεπε να δούμε περισσότερα τέτοια παραδείγματα, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Φρεντ Νόιμαν που θα μας το παρουσιάσει αυτό. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Πρόεδρο που μας ε, δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αυτό το νέο ε, πρόγραμμα για νέους, DotWise, το οποίο επικεντρώνεται σε δύο από τα σημαντικά θέματα της έκθεσης, τα νέα μέσα ενημέρωσης και τους νέους. Οι νέοι δεν αναγνωρίζουν την παραδοσιακή ε, πολιτική ε, ε, επικοινωνία και πληροφόρηση και γι' αυτό σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τους νέους για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους ηλικιακή ομάδα 25 με 25 ετών αποτελούν το 20% του ε, πληθυσμού της Ευρώπης. Ε, αυτά είναι τα ε, εκατομμύρια για τα οποία μιλάει η Επιτροπή στην έκθεσή της. Λέει ότι λιγότερο από το 40% των νέων ηλικίας 16 με 29 ετών εμπιστεύονται τους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 60% των νέων της Ευρώπης δεν πιστεύει τους πολιτικούς, δεν πιστεύει στους πολιτικούς και στα πολιτικά κόμματα. Όταν λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια πολιτική κοινότητα που να βασίζεται στην ε, ε, πολυμορφία μας, οι νέοι ήδη μας έχουν εγκαταλείψει. Οι νέοι θέλουν να αναπτύξουν την ε, ισότητά τους και την πολυμορφία τους σε άλλο επίπεδο, σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα. Η Ευρώπη των νέων δεν είναι ταυτόσιμη με την ε, Ευρώπη των πολιτικών. Υπάρχει ένας ε, ψηφιακός ε, κόσμος ο οποίος δεν καθοδηγείται από τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά από τις δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων. 250.000 νέοι χρήστες εμφανίζονται κάθε μέρα στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι δηλαδή ένας κόσμος σε ραχταία ανάπτυξη. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς άλλο μέσο ενημέρωση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στον ίδιο ρυθμό. Για παράδειγμα, για την τηλεόραση χρειάστηκαν 13 χρόνια για να ε, έχουν 50 εκατομμύρια θεατές, ενώ το Facebook πέτυχε να έχει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες σε λιγότερο από 9 μήνες. Πάνω από 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν ε, τα κοινωνικά μέσα όπως είναι το Facebook, το YouTube και το Twitter. Και αναμένεται το νούμερο αυτό να ξεπεράσει τα 107 εκατομμύρια μέχρι το τέλος ε, του 2012. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για ευρωπαϊκή και παγκόσμια τροποποίηση των συνηθιών μας όσον αφορά τα μέσα ενημέρωση, αλλά και αλλαγή της κατανάλωσης μιας γενιάς ε, των μέσων ενημέρωση, και, καθώς και ε, τροποποίηση του τρόπου επικοινωνία των νέων. Ήδη σε ηλικία 5 ετών πάνω από το 40% των ε, νέων ε, καταχωρούνται ως ε, χρήστες, μόνιμοι χρήστες του διαδικτύου, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίε χρησιμοποιούν οι νέοι κάθε μέρα το διαδίκτυο. Κάνουν surfing, κάνουν chat και οι δραστηριότητες που βασίζονται στο διάλογο αποτελούν σημαντικό κομμάτι το, της ζωής των νέων. πάρα πολλά εκατομμύρια νέοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα και πάνω από τους μισούς από ε, επικαιροποιούν συνέχεια το προφίλ τους. Και τι κάνουν εδώ, έχουν επαφέ με τους φίλους τους, ε, επεκτείνουν τον ε, κύκλο νέων, ε, ανταλλάσσουν ε, επεκτείνουν την κοινωνική τους ζωή χωρίς κοινωνικές και χωρίς κοινωνικούς και εθνικούς περιορισμούς. Ε, τα κοινωνικά μέσα μπορούν να ε, μαγνητήσουν και να διατηρήσουν την ε, επαφή των νέων. Μπορούν εδώ να έχουν επαφή μεταξύ τους οι νέοι και οι νέοι παρουσιάζουν στιγμιότυπα της ζωής τους που δείχνουν την πολυμορφία της γενιάς αυτής, από την άλλη περιγράφουν και τα, τις ομοιότητες των νέων με βάση την ε, κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητά του, είτε, ε, είτε το συνειδητοποιούν αυτό οι νέοι είτε όχι. Ακριβώ αυτά τα στοιχεία ε, είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμεί στο πρόγραμμά μας. Δημιουργούμε ένα φόρουμ κινηματογραφικό όπου οι νέοι μπορούν να επιδείξουν αλληλεγγύη σε διασυνοριακό επίπεδο. Με άλλα λόγια, δημιουργούμε Ε, έναν χώρο για την, για την νεολαία της Ευρώπης, ε, η οποία από την ε, διαφοροποίησή της, την πολυμορφία της, αλλά και την κοινωνική της ταυτότητα. Το DocsWise έχει να κάνει με την αφήγηση ιστοριών από νέους προς νέους. Τη δουλειά την κάνουν νέοι κινηματογραφιστές και πολύ πρακτικά γίνεται το εξής Τέσσερις νέοι σε κάθε χώρα λαμβάνουν μια ε, κάμερα και ε, όπως και σε ένα ημερολόγιο μας μιλάνε για τη ζωή τους, ε, για τα προγράμματά τους, για τις επιλογές τους, για τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν, που είναι τα πάντα για αυτούς στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όλοι αυτοί έχουν την αίσθηση ότι είναι μοναδικοί, ότι είναι πρωτότυποι, ότι αντιμετωπίζουν μόνοι τους το σημαντικό τους πρόβλημα, τις εσωτερικές τους σκέψεις, την λήψη αποφάσεων τους κλπ. Πολύ λίγοι από εμά όμως είμαστε μοναδικοί, διότι ε, έτσι φαίνεται ότι και άλλοι νέοι συμμερίζονται τις ίδιες σκέψεις, ε, την ίδια οπτική και ακριβώς εδώ υπάρχει μοναδική ε, ευκαιρία για τους νέους να ε, να πετύχουν την αναγνώριση των προβλημάτων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι νέοι αυτοί ε, αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα ε, που είναι πιο πραγματική από αυτή που βλέπουμε στα ε, παραδοσιακά μέσα ενημέρωση. Διότι όταν οι νέοι μπορούν να διαχειρίζονται τη δική τους πλατφόρμα, ε, δημιουργείται μια διάδραση ανάμεσα στους χρήστες που βασίζεται ε, στον σεβασμό, στην περιέργεια και στο ενδιαφέρον που έχει ο ένας για τον άλλον. Το DocsWise δεν είναι πολιτική επικοινωνία, ούτε είναι προσπάθεια ε, να χρήσεις μιας πολιτικής ατζέντα στους νέους, διότι αυτό, πιστέψτε με, θα το καταλαβαίναν αμέσω οι νέοι και θα εξαφανίζονταν από την πλατφόρμα αυτή. Το DocsWise είναι ένα μέσο για να ε, επικοινωνήσουμε όσον αφορά τις αξίες των νέων. Εάν θέλουμε να προωθήσουμε κοινή κατανόηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, θα πρέπει να δώσουμε στους νέους έναν χώρο όπου θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν την προσωπική τους και εθνική συνείδηση και θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επικοινωνήσουν ε, πέρα από τα εθνικά και γεωγραφικά σύνορα για να δημιουργήσουν κοινέ εμπειρίες. Και πιστέψτε με, οι νέοι τη Ευρώπης έχουν πολλές καλές ιστορίες οι οποίες προκαλούν έκπληξη, ε, συγκλονίζουν, αλλά ε, βασίζονται στην επιθυμία διαλόγου μιας ολόκληρης γενιάς. Στην Δανία το 2008 και 2009 ε, εφαρμόσαμε ως πιλωτικό πρόγραμμα το DocsWise ε, κάθε φορά με τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάστηκαν από κάποιον νέον κινηματογραφιστή ντοκιμαντέρ. Είχαμε για παράδειγμα 18χρονο νέο από την Ήπεθρο που ε, ανεξαρτητοποιόταν από τους ε, γονείς του και έπρεπε να δημιουργήσει το δικό του σπίτι. Μία ε, λεσβία 22 ετών που ήθελε να ε, συνδυάσει τις δικές της φιλοδοξίες για το μέλλον της ε, και με το πρόβλημα ότι μια μεγάλη πόλη δημιουργεί πολλές, ε, ε, πολλούς πειρασμούς, ε, πολλά πάρτι, αλκοόλ κτλ. Έναν άλλο νέο είχαμε που θα πήγαινε στο Αφγανιστάν. Επί 10 εβδομάδες παρακολουθήσαμε την, τον αποχαιρετισμό του από την οικογένειά του για να πάει στον πόλεμο και επίσης ε, έναν ε, νέο που περιγράφει την, ε, το διχασμό ανάμεσα στην Δανέζικη και την Ισλαμική κοινωνία και που έφερε άλλους νέους μέσα στο σπίτι του για να δουν ακριβώς τα προβλήματα αυτά. Θα ήθελα να σας δείξω κάποιες από τις ταινίες αυτές για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάω και να θυμάστε Κανένας άλλος εκτός από τους νέους δεν αποφασίζει τι θα δείξει η κάμερα ή τι θα πει η ιστορία τους.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 Øh, Ζητώ συγγνώμη που υπήρχε μια καθυστέρηση ε, ανάμεσα στο κείμενο και στον ήχο. Ε, το πρόγραμμα DocsWise ε, είναι σχετικά απλό και είχε μεγάλη επιτυχία στη Δανία. Θα θέλαμε τώρα να παρουσιάσουμε ε, στους νέους της Ευρώπης την ευρωπαϊκή εκδοχή. Στην ευρωπαϊκή εκδοχή του DocsWise, docswise.eu, προτείνουμε πιλωτικό πρόγραμμα με 4-5 συμμετέχουσες χώρες και με 4 νέους συμμετέχοντες σε κάθε χώρο. Δηλαδή 16 με 20 νέους οι οποίοι ε, σε ένα, για κάποιο χρονικό διάστημα θα κινηματογραφούν τη ζωή τους ε, και θα περιγράφουν τις ε, αποφάσεις ε, που αντιμετωπίζουν. Στην Δανία, στην κάθε χώρα, επιλέγεται ένας που θα κινηματογραφεί και σε κάθε μέρα θα δημοσιεύεται ένα νέο κομμάτι και θα μπορούν οι χρήστες να σχολιάζουν στο διαδίκτυο τις συνεισφορές. Το docswise.eu αναπτύσσει του, τις λειτουργίες δηλαδή που ήδη υπάρχουν στο YouTube και στο Facebook. Δεν θα μιλάμε απλά για μικρές ταινιούλες, αλλά για μια συνεχή κινηματογραφική ιστορία με μια επιλογή νέων από την Ευρώπη. Και δεν θα έχουμε απλά ε, αδιάφορες ε, ε, περιγραφές, θα μιλάμε για ε, συναισθήματα και σκέψεις των νέων που θα μεταφέρονται κινηματογραφικά και εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορούν να ε, τα βλέπουν αυτά στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύουμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή πολιτική επικοινωνία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει τρόπος ε, να επικοινωνήσουμε, ε, να παρουσιάσουμε την πολυμορφία μας και τις αξίες μας απέναντι στους νέους. Και πιστεύουμε ότι με το πρόγραμμα DocsWise EU θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διάλογο μεταξύ των νέων και να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα και την επιθυμία να συζητήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και την Επιτροπή που ε, μας ακούσατε και ελπίζω να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο κόσμο μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Φρέντι Νόιμαν για την παρουσίαση αυτή και που μας έδειξε ένα παράδειγμα του τι μορφή μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, ποια είναι η πραγματικότητα που θα μπορούμε να έχουμε εάν τολμήσουμε να αφήσουμε ε, κάποιον ε, να ε, μπει στο χώρο μας που να έχει επικοινωνία με τους νέους. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το τελευταίο σημείο της έκθεσής μου έχει να κάνει με την αφήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας, διότι όπως είπε ήδη στις δηλώσεις της για το θέμα αυτό, το θέμα εδώ είναι να αφηγηθούμε μια ιστορία. Και βέβαια τίθεται το ερώτημα ποια ιστορία. Τα τελευταία 50 χρόνια η ιστορία πάντα ήταν ότι πρόκειται για ένα ε, εγχείρημα το οποίο έχει να κάνει με την ειρήνη, την ε, ευημερία και τη δημιουργία μιας κοινωνίας στην Ευρώπη ε, για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Και είναι πολύ ωραία η ιστορία αυτή, αλλά πιστεύω ότι οι νέοι της Ευρώπης, οι νέοι που μεγαλώνουν σήμερα στην Ευρώπη έχουν συνηθίσει το έχουν συνηθίσει αυτό, το οποίο σημαίνει ότι καλός ή κακός θα πρέπει να καλό η κακό θα πρεπει να προχωράει ακόμα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό χρειαζόμαστε χρειάζεται να, να ανανεώσουμε το όραμά μας, να το πω έτσι. Ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το νέο όραμα και να το αφηγηθούμε με τους τρόπους αυτούς. Και θα ήθελα να πω ότι παντού στο σύστημα και μεταξύ άλλων και εμείς οι βουλευτές εκπαιδευόμαστε στο θέμα της επικοινωνίας, διότι παρότι όλοι, είπα ότι όλοι είμαστε ε, ειδικοί στην επικοινωνία, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και είναι σημαντικό για τους υπαλλήλου και για τους πολιτικούς να μπορούν να επικοινωνήσουν. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ τον εισηγητή και τον δανό εμπειρογνώμονα. Ε, ήταν ε, πολύ επίκαιρο και νομίζω ότι όντως ε, συνειδητοποιεί κανείς όταν βλέπει κάτι τέτοιο ότι υπάρχουν δυνατότητες να στηρίξουμε μία προσπάθεια εδώ. Ο Βιμ Βέντερς, ο μεγάλος σκηνοθέτης, είχε πει στο Βερολίνο πριν δύο-τρία χρόνια στις τελευταίες, στους τελευταίους αιώνες έχουμε παραλείψει να εξηγούμε τις ευρωπαϊκές ιστορίες. Πάντοτε καταναλώναμε αυτά που μας έλεγε η Αμερική ενώ τις ιστορίες μας από την Πορτογαλία ως την Εστονία δεν τις έχουμε εξηγήσει. Είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει ε, να λάβουμε σοβαρά. Η εξιστόρηση αυτή είναι σημαντική. Ε, θα πρέπει τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να παρακολουθήσουν. Υπάρχει μία νέα εποχή της επικοινωνίας επικοινωνίας και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που καταφέρετε να τα κάνετε αυτά με τόσο ενθουσιασμό και τόσα μέσα. Ε, πρόκειται ε, για εκθέσεις κατά πρωτοβουλία τις οποίες μπορούμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, να τους εξηγήσουμε τι έχει γίνει ήδη. Έχω έξι συναδέλφους οι οποίοι έχουν ζητήσει τον λόγο. Καταρχήν ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας που έθεσε προς συζήτηση αυτό το πρόβλημα της απόλυτης καταστροφής της ε, πληροφόρησης και επικοινωνίας των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι ο μόνος τομέας που τα τελευταία 30 χρόνια, αν το παρακολουθήσουμε, βλέπουμε να οπισθοχωρεί συστηματικά. Αυτό όμως δεν ανησυχεί τους Ευρωπαίους ηθήνοντες από ό,τι φαίνεται. Όπως γνωρίζετε ορισμένοι, έχω τη διπλή εμπειρία να είμαι ευρωβουλευτής. Είναι η δεύτερη μου θητεία βέβαια, άλλοι θα έχετε παραπάνω φυσικά. Αλλά από την άλλη μεριά ήμουνα δημοσιογράφος στη χώρα μου και ήμουνα και ιδιοκτήτης ΜΜΕ και πάντα εκπληζόμουν από αυτήν την τεράστια αλαζονία με την οποία τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, ασκούν αυτή την πολιτική της πληροφόρησης, εκφράζονται, δεν εκφράζονται. Σας ευχαριστώ κύριε Λόγκεγαρτ που τονίσατε αυτή την έλλειψη ορατότητας των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Πραγματικά βάλατε το δάχτυλο στην, στην πληγή. Ξέρετε, έχουμε εμείς αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία τελικά είναι οριζόντια δίκτυα Συζήτηση και είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή. Αυτό είναι ένα βέβαια από τα σημεία, αλλά δεν είναι το μόνο. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να πω ότι είναι εκπληκτικό εκπληκτικό το ότι η Κομισιόν δεν κατάφερε να μας φέρει κοντά αυτό το, αυτή τη μερίδα των εφήβων 14-16 ετών που είναι πάμπολοι σε όλη την Ευρώπη. Και για την Ευρώπη δεν υπάρχει τίποτα στα βιβλία ιστορίας, αν δεν υπάρχουν δυο σελίδες όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες σελίδων σε θέματα μαχών, βαρβαροτήτων, κρυμάτων. Οι νέοι 13-14 ετών στη Γαλλία έχουν ένα βιβλίο ιστορίας με δύο σελίδες για την Ευρώπη και 250 για τα υπόλοιπα. Και το γεγονός ότι η χώρα μου, η Γαλλία, έχει ως α την εθνική ταυτότητα και ως β την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δεν βρίσκονται πουθενά, δεν αντικατοπτρίζονται πουθενά αυτά. Οι χώρες έχουν τεράστιες ευθύνες. Εδώ και 20 χρόνια σχεδόν δεν ακούω να συζητείτε στην Ευρώπη η ευρωπαϊκή οικοδόμηση, που σήμερα είναι εντάξει, ευρωπαϊκή στασιμότητα, και εγώ αυτά τα λέω πολύ καθαρά, ξέρετε. Λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη αφού τα έχω σκεφτεί πρώτα. Λοιπόν, βλέπω την Ευρώπη από τη μια να είναι ένα χρήματο κυβότιο όπου μια κυβέρνηση προσφεύγει και παίρνει χρήματα από αυτό το χρήματο κυβότιο, αντί για τους φορτηγατζίδες, για τους ψαράδες κτλ. Και γυρίζει πίσω στη χώρα του και λέει ορίστε με αυτά τα λεφτά στο χέρι, λέγοντας εγώ σας υπερασπίστηκα, λες και εδώ στις Βρυξέλλες ήταν ένα κέντρο διεθνών επιθέσεων. Και τι γίνεται. Σε δεύτερη φάση μιλούν αρνητικά όταν ένα μέτρο αποφασίζεται σαν να είναι ένας μεθυσμένος χωροφύλακας ο οποίος παίρνει αποφάσεις χωρίς να τις δικαιολογεί μόνο και μόνο για να πλήττει τους λαούς. Ο Ελί Βίζελ τι λέει, Λέει με την περίφημη φράση, πάνω κάτω τη λέω, λέει ο μιλητής, μια χώρα που δεν γνωρίζει την ιστορία της, οι νέοι που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους, ρισκάρουν να ξαναζήσουν αυτή την ιστορία. Εμείς στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες, φέρουμε τεράστιες ευθύνες. Το είπα και το ξαναείπα στον ε, πρόεδρο της τωρινής επιτροπής, είδατε βέβαια τη χρήση που έκανε, όλοι τη βλέπετε ότι υπάρχουν μερικά ελαττώματα και μορφολογικού χαρακτήρα πολλές φορές βέβαια και επί της ουσίας. Ας δούμε λοιπόν πρώτα την ουσία. Οι συζητήσεις δεν είναι ιεραρχημένες. Πώς θέλετε οι πολίτες να κατανοήσουν πώς είμαστε, πόσο χρήσιμοι είμαστε για τους λαούς όταν η πιο βαριά κρίση που γνωρίζουμε από το 29 και μετά δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης. Ποια είναι η ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτή την κρίση. Κύριε Λόγκεγκαρτ, εμεί δεν μπορούμε να, ασκούμε καλή επικοινωνία εν απουσία πολιτικής και στην προκειμένη κρίση δεν υπάρχει πολιτική. Γίνονται απόπειρες εναρμόνισης κοινή εναρμόνιση ορισμένων στοιχείων που είναι καθαρά εθνικού χαρακτήρα. Αλλά να σταθώ σε ένα άλλο σημείο να αφήσω την κρίση. Πέντε-έξι χρόνια δεν ακούω να μιλιέται αυτό εγώ εδώ στο Κοινοβούλιο και συντόρι σίγουρα πολλά παραπάνω. Λοιπόν έρευνα, ευρωπαϊκή έρευνα, ακούσατε εσείς και δεν ακούγεται. Υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες, ε, ερευνητές αριστερά, δεξιά, ανά τον κόσμο. Ακούσατε ποτέ τίποτα. Και αυτό γιατί. Διότι αντί να καταφέρουμε να έχουμε μία δανειοδότηση θεάς ουσίες για τη χρηματοδότηση αυτών των ερευνητών που φεύγουν στη Δυτική Ακτή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγοι στην Βρετανία και τώρα έχουν αρχίσει και διαραίουν οι εγκέφαλοί μας στην Κίνα. Δεν έχουμε καμία πολιτική, συζητιότανε κάποτε για αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε ότι σε όλη αυτή την οχέλεια υπάρχει και, μία, και ένας απόϊχος του 1937. Ακούω εγώ να γίνεται συζήτηση για την Ελλάδα. Πολλά λέγονται. Αλλά εσείς ακούσατε ποτέ μία οικογένεια όπου ένα μέλος της είναι άρρωστο και το πετάνε από το φορτηγό, το πετάνε από το βαγόνι, το πετάνε από το, το δωμάτιο, το πετάνε από από το σπίτι. Μα αυτό δεν γίνεται. Βλέπετε λοιπόν τη, μικρο, μικροψυχία για τα ελληνικά πράγματα. Και τι αποδεικνύουμε εμείς σε όλους τους κερδοσκόπους αποδεικνύουμε ότι έχουν μακροημέρευση μπροστά τους. Διότι εμείς κάνουμε μια τιτίζικη πολιτική. Ξεψυρίζουμε και αύριο οι ιστορικοί θα το θυμούνται αυτό. Λοιπόν, εντάξει, προσγειώνομαι, προσγειώνομαι. Εγώ θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι επαρκώς διαφανή. Φτάνει το κοινοβούλιο να, πούν, να πει ορισμένα πράγματα. Οι δημοσιογράφοι είναι πανταχού παρόντες στους διαδρόμους και είναι... και έχουν στη διάθεσή τους όλη την πληροφόρηση. Πολύ λιγότερο η Κομισιόν βέβαια, πολύ λιγότερο το Συμβούλιο. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε πολιτισμό της εικόνας και σε αυτό δεν έχουμε καμία σύσταση. Εγώ είχα πει στην Κομισιόν να αφαιρέσει την Παρασκευή από την ατζέντα της και να στέλνει τους επιτρόπους σπίτια τους. Να τους στέλνει, αν όχι στα σπίτια τους δηλαδή, να τους στέλνει στις όμορες χώρες του Βελγίου και να λένε στον κόσμο δέστε τι κάναμε αυτή τη βδομάδα, δέστε ποια ήταν η δράση μας, ακούστε. Ήταν επανευτυχής ο πρόεδρος της Κομισιόν από αυτή την ιδέα, είδατε τι απόγεινε. Για να έχουμε λοιπόν επαφή επικοινωνίας με τον κόσμο πρέπει να έχουμε ουσία και όχι αξεσουάρ και πρέπει να έχουμε καθαρό λόγο για να μιλούμε στο λαό. Ευχαριστώ τον κύριο Καβαντά. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους επόμενους συναδέλφους να μην ε, μακρηγορούν τόσο πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αλλά είναι λιγάκι πιο γρήγοροι. Ε, κύριε Καβαδά, έχει το λόγο, ζητώ συγγνώμη. Η επόμενη μειοελήτρια. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρωτοβουλία αυτής της έκθεσης και πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος επικοινωνίας και να προωθηθεί με κάθε τρόπο, διότι υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ήδη αναφέρατε και επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αναφέρομαι εις ε, την ε, προώθηση της ε, επιμορφώσεως των δημοσιογράφων, τα μέτρα που μπορούμε να βελτιώσουμε σαν Κοινοβούλιο ή σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εν πάση περιπτώσει, στην έκθεση αυτή έχω διάφορα προβλήματα και δεν τα αποσιωπώ. Δεν έχω ο, <clears throat> καμία αντίρρηση να υπάρξει μία έκκληση ε, για να ε, προωθηθεί το θέμα αυτό στα ευρωπαϊκά μέσα Αλλά αν κοιτάξουμε τους δημοσιογράφους ε, στις Βρυξέλλες και διαπιστώσουμε ότι όλο και περισσότεροι ανταποκριτές μειώνονται και δεν είναι τα δημόσια μέσα τα οποία αποσύρουν τους ε, δημοσιογράφους αλλά τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης που δεν ε, οργανώνουν πλέον παραγωγές τότε θα πρέπει να απευθύνουμε τις εκκλήσεις μας όχι μόνο στα δημόσια μέσα ενημέρωσης αλλά και στα ιδιωτικά ε, διότι βλέπουμε ότι μειώνται συνεχώς οι ανταποκριτές στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι στην έκθεση σε διάφορα σημεία υπάρχει ε, μία μια ε, αποσιοποίηση της κατανομής των ε, αρμοδιοτήτων διότι βλέπουμε ότι ε, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, μπορεί να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διόρθωσή τους. Αυτό φαίνεται ίσως περιορισμένο, περιορισμένης εμβέλειας, αλλά ουσιαστικά δεν πρέπει να θίξουμε την ελευθερία του τύπου και της αναμεταδόσεως. Δηλαδή έχουμε αγαθά τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε στην Ευρώπη και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ε, διότι αυτή η ε, στενοπός ε, η οποία τονίζεται ιδιαίτερα στη Γερμανία συνταγματικά δεν πρέπει να κλείσει. Επίσης πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα κάθε χρόνο αξιολογεί τα προγράμματά της όσον αφορά την ευρωπαϊκή πτυχή αλλά και εδώ δεν πρέπει να υπερβούμε τα όρια όσον αφορά τον ε, έλεγχο της ε, κρατικής ε, ραδιοφωνίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ διότι αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν εκτελεστικό όργανο για την κατανομή των αρμοδιοτήτων δεν είναι κατάλληλη για να προβεί στον έλεγχο αυτών γιατί θα πρέπει η ελευθερία του ραδιοφώνου να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών. Επίσης ε, δεν συμφωνώ την προώθηση της άμεσης ε, χρηματοδότησης περιοδικών ε, που ε, δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει και εδώ να προσέξουμε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν πρέπει να θίξουμε την ελευθερία του τύπου διότι δεν είναι προς όφελος κανενός να ε, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δικά της περιοδικά για να προωθούν μια συγκεκριμένη εικόνα της Ευρώπης. Ούτε εσείς το θέλετε κύριε Λόκεργκαρ αλλά υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο διαγράφεται σε ορισμένα σημεία της έκθεσης αυτής και θα επιθυμούσα σε ορισμένα σημεία από κοινού να ξανακοιτάξουμε τι γίνεται για να υπάρξουν σαφείς ε, ε, διαχωρισμοί μεταξύ ε, της ε, ελευθερίας της συντακτικής και της δημοσιεύσεως και σε διάφορα παρεμφερή θέματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ήβεν. Υπάρχει ανταγωνισμός ε, Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ και μεταξύ των δημοσίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η δραστηριότητά μας να ανανεωθεί Θα πρέπει να είμαστε εύστοχοι, να έχουμε νέα πιο ζωντανά, ούτως ώστε τα ιδιωτικά ΜΜΕ να ασχοληθούν μαζί μας. Ξέρουμε επίσης ότι όσοι ενδιαφέρονται για τις ειδήσει, ενδιαφέρονται περισσότερο για τις τοπικές ειδήσει και όχι για τις διεθνείς ειδήσει. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς ε, να μετατρέψουμε αυτές τις ειδήσει σε ειδήσει ενδιαφέρουσες, ούτω ώστε και σε τοπικό επίπεδο να ενδιαφέρουν το πολίτη, όχι μόνο διεθνώς. Κυρία Βιλανόβα. Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι πρόκειτο για μία στρατηγική επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όχι μία νέα στρατηγική και θα ήθελα να δεχθούμε τη δυνατότητα τροπολογιών διότι αυτό που παρουσιάζεται τονίζει περισσότερο τα νέα μέσα ενημέρωσης ε, που αναφέρονται σε δύο σημεία αλλά θα έπρεπε να επεκταθούμε περαιτέρω όχι για την ύπαρξη αυτών των νέων μέσων αλλά και το θέμα της ασφαλείας στο διαδίκτυο διότι έχουμε ε, ε, αναφέρει ότι 52% των ε, παιδιών μικρής ηλικίας είναι εγγεγραμμένα στο διαδίκτυο και Πρέπει να προσέξουμε πώς μπορεί να επηρεαστεί η παιδεία τους. Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένε τροπολογίες όπου θα τονίζουμε ότι τα νέα μέσα ενημέρωσης είναι χρήσιμα, έχουν συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορέσαμε πολλά περιστατικά <clears throat> να τα συζητήσουμε πολύ γρήγορα με αυτά τα νέα μέσα, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Ο Ιβο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι πολύ, η έκθεση, είναι πολύ καλή η έκθεση του κυρίου Λεκεγκάρτ. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως είπατε και όπως είπε και ο κύριος Καβαντά. Ήμουν δημοσιογράφος σε δημόσιο κανάλι και ξέρω πόσο σημαντικό είναι το θέμα και πιστεύω ότι πράγματι θα πρέπει να έχουμε ένα scoreboard, ένα πίνακα αποτελεσμάτων για να μπορέσουμε να σπρώξουμε τα δημόσια κανάλια προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Ο κύριος Καβαντά έχει επίσης δίκιο. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να εξετάσουμε προσεκτικά την παράγραφο 5. Επίσης έχει δίκιο η κυρία Νεβιτάλοβα ε, που λέει ότι ναι, πρέπει να τα πετύχουμε αυτά. Πώς θα τα πετύχουμε όμως. Έχουμε έναν αριθμό δημοσιογράφων και ανταποκριτών στις Βρυξέλλες και Αυτοί καλύπτουν ε, την κατάσταση, αλλά τα νέα μέσα αναπτύσσονται πάρα πολύ ε, γρήγορα. Ε, βλέπουμε και ότι οι συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου ε, εκπέμπονται στο διαδίκτυο. Έτσι, πολλοί δημοσιογράφοι μπορούν να τα παρακολουθούν αυτά από το λάπτοπ τους. Δεν χρειάζεται να έρθουν στις Βρυξέλλες. Αυτά που είπατε για την παιδεία είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει οι ευρωπαϊκές υποθέσεις να αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πριν την τελική ψηφοφορία για την έκθεσή σας. Ίσως να μπορούσαμε να έχουμε μια μελέτη σχετικά με την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Ξέρω περίπου πώς έχει η κατάσταση στα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Και έχω κάποιες ερωτήσεις. Στην παράγραφο 17 αναφέρεστε στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρεστε σε μια επιχειρησιακή ομάδα που θα απαρτίζεται από ανεξάρτητους δημοσιογράφους. Έχω κάποιες επιφυλάξεις. Δεν ξέρω ποιος θα το πληρώσει αυτό, ποιος θα το χρηματοδοτήσει αυτό. Μήπως έτσι ανταγωνιζόμαστε τα υπάρχοντα μέσα ενημέρωσης, τα τυπωμένα και τα επιγραμμικά, όπως το EU Observer ή την European Voice και άλλα. Ίσως θα ήταν καλύτερο να συνεργαστούμε με αυτά, να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πιο δημοφιλή και πιο ανοιχτά απέναντι, πιο προσβάσιμα από το ευρύ κοινό. Πώς το βλέπετε αυτό, ίσως θα ήταν άλλος τρόπος να πετύχουμε τον ίδιο στόχο. Και μία τελική ερώτηση για την παράγραφο 23. Αναφέρεστε στην δημιουργία επιγραμμικών φόρουμ όπου οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Θα μπορούσαμε ίσως να δημιουργήσουμε ένα επιγραμμικό φόρουμ θα είναι καλό μέσο αυτό και για τα σχολεία, θα ήταν ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάτι τέτοιο. Και μια ερώτηση που συνδέεται με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι το δικό μου θέμα. Τι, κάνει, τι κάνουν τα κανάλια και τι κάνει ο, ο τύπος μέσω των ιστοσελίδων τους. Μπορεί να υπάρχει εδώ ανταγωνισμός θα μπορούσαμε ενδεχομένως ε, να έχουμε ένα καλό επιγραμμικό φόρουμ μέσω των ιστοσελίδων των εφημερίδων. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε πέντε που έχουν ζητήσει το λόγο ακόμα. Έχουμε ακόμα μία ε, έκθεση και έχουμε τον συνάδελφο Μαρτίνες Μαρτίνες. Παρακαλώ όλους τους συναδέρφους να περιοριστούν στο 1,5 λεπτό ώστε να προλάβουμε και την επόμενη έκθεση του Ιβο Μπέλετ για τα μέσα ενημέρωση. Είμαι λίγο αγενή τώρα, διότι άφησα να, μιλήσετε αρκετά, αλλά δίνω το λόγο στον συνάδελφο. Κοιτάστε, εγώ είμαι κάπως σκεπτικιστής ε, ως ε, προς την παρουσίαση του προλελήσαντος <coughs> και η παρουσίαση του επικύρωσε τον σκεπτικισμό μου. Εγώ θεωρώ ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι οι πολιτικοί να αρχίσουν να ρυθμίζουν τα ΜΜΕ. Ε, εμείς έχουμε εμπειρία στις διάφορες χώρες στα εθνικά κοινοβούλια σχετικά. αν εμείς πρέπει να ρυθμίσουμε αυτού του είδους τη δουλειά, τότε τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να ρυθμίσουν. Και σε τελευταία ανάλυση, δεν είμαστε εμείς που κρίνουμε τους δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι κρίνουν εμάς. Αν εμείς είμαστε απόντες, από τα ΜΜΕ γιατί κάνουμε πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, φυσικά δεν ενδιαφέρονται και για μας. Αν για 20 λεπτά καθόμαστε και μακρηγορούμε αερολογώντας και μετά σκονόμαστε και φεύγουμε, μα φυσικά δεν ενδιαφέρονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μας. Ελεύθερη να πρέπει να είναι τα ΜΜΕ. Και η πολιτική είναι η τελευταία ομάδα η οποία θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται τα ΜΜΕ. Αν εμείς ε, θεωρούμε ότι τα, η αγορά της επικοινωνίας είναι τέτοια που θα πρέπει να ασχοληθεί με τη δική μας δουλειά, αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να το έχουν άλλοι και όχι εμείς. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ τον κύριο Λόκεργαρτ για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι αυτά που αναφέρονται είναι ε, καλά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πολλά από αυτά δεν θα μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στην πράξη. Διότι ξέρουμε ε, ότι προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να επικοινωνήσουμε για το τι συμβαίνει και πρόκειται για έναν περίπλοκο θεσμικό έργανο, τα κράτη-μέλη λειτουργούν διαφορετικά διότι ο Βρετανικός τύπος είναι ο πλέον ευρωσκεπτιστικός. Παρόλο λοιπόν που δεν διαφωνώ θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι μία ε, μέθοδος η οποία αποδίδει υποχρεωτικά. Υπάρχουν δυνατότητες βελτιώσεως. Θέλω λοιπόν ε, να πω ότι έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό επί ετών και για να έχουμε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κάλυψη στα κράτη-μέλη θα το επιτύχουμε μόνο εάν επικοινωνούμε με τους δημοσιογράφους στα κράτη-μέλη διότι οι Βρετανοί δημοσιογράφοι πλην του BBC ε, δεν ακούνε κανέναν άλλον και αν ε, τον ακούσουν θα είναι μόνο αρνητικά και οι ε, δημοσιογράφοι δεν συμφωνούν υποχρεωτικά με το δικό μας πρόγραμμα οπότε υπάρχουν θέματα τα οποία θέλουμε να προβάλλουμε και μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα αλλά όπως Είπατε πολύ σωστά, αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κρατών μελών και ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέψει να ε, επικοινωνήσουμε αμέσως με τους δημοσιογράφους και αυτό είναι που πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ρόβεκερ, διότι έχει συντάξει μια έκθεση πολύ σημαντική, επικέντρωσε επικέντρωσε την προσοχή του σε ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που έχουμε, δηλαδή το πώς εμείς πρέπει να φέρουμε προς τα έξω την Ευρώπη. Εμείς έχουμε δύο προβλήματα για τα οποία πολλές φορές η Ευρώπη δεν γίνεται αντιληπτή. Καταρχήν πολιτικά, διότι πολλές από τις αποφάσεις που πρέπει να γίνουν πρώτα αντιληπτές από τις ίδιες τις εθνικές αρχές. Και οι εθνικές αρχές όταν μεταφέρουν αυτό το μέτρο το κοινοτικό, ε, τη συζήτηση την καθιστούν εθνική. Και όταν δίνονται τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, περνάνε η χρηματοδότηση πάλι από ε, από τα τοπικά. Όργανα. Είναι οι περιφέρειες οι οποίες μοιράζουν τη χρηματοδότηση. Τώρα, οι νέοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Ξέρουν πολύ καλά ποια είναι τα σύνορα ότι δεν είναι πια τα εθνικά σύνορα, δεν είναι τα τοπικά σύνορα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε εμεί τον τρόπο να προσελκύσουμε το κοινό. Αλλά πρέπει να βρούμε και κάτι ενδιαφέρον. Και ό,τι εκπομπές γίνονται γύρω από την Ευρώπη, γενικώ θα τις παρακολουθεί κανένας γιατί είναι βαρετές. Πρέπει να βρούμε λοιπόν κάτι πιο ενδιαφέρον για να ενημερώνει το κόσμο για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριε... Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεβαλτ γιατί έθεσε θέματα πολύ βασικά. Υπάρχει το θέμα του πλουραλισμού και της ελευθερίας των ΜΜΕ όπως επίσης και οι εθνικοί εθνικές αρμοδιότητες είναι ένα θέμα που τίθεται και μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή να τεθούν οι βάσεις στα ΜΜΕ ούτως ώστε η ευρωπαϊκή ηθαγένεια να γίνει ενεργή ηθαγένεια τα διάφορα μέσα που υπάρχει στη διάθεσή του ο ευρωπαϊκός λαός να είναι δικαιώματα απαιτούμενα, εφαρμοζόμενα. Δεν είναι λάθος λοιπόν αυτό. Δεύτερο, η εμπειρία που μας δείξατε είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πιστεύω ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να προθήσει ακροάσεις παρουσιάσεις για να δημιουργηθούν κίνητρα και ένα νέο πρόγραμμα ίσως που θα μπορούσαμε να προτείνουμε για να υποστηρίξουμε κοινωνικές πλατφόρμες, ε, media, που να είναι πιο ενεργητικό, πιο ενδυναμωτικό για την Ευρώπη. Τώρα για το δημόσιο ιδιωτικό σύστημα media. Στη χώρα μου υπάρχουν μέσα, όπως και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, όταν δίνεται η παραχώρηση των διαφόρων ζωνών του εθέρος, που είναι κοινό αγαθό, να θέτουμε όρους. Να θέτουμε, ας πούμε, τον όρο της υποχρέωσης πληροφόρησης σε ορισμένα περιεχόμενα, όχι ως λογοκλησία, πρόθεση. Αυτό είναι ένα σημείο. Και σε εθνικό επίπεδο να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα κοινοτικά θέματα. Εμείς αυτό το παλεύουμε στη χώρα μας, διότι υπάρχει μια μεγάλη αδιαφορία, ουσιαστικότατη αδιαφορία γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα. Πρώτο ζήτημα. Πώς να πληροφορούμεθα αποτελεσματικά για τα πιο ουσιαστικά θέματα. Και κυρίως για ό,τι έχει επιπτώσει στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε στη συνεργασία, με τα εθνικά δημόσια μη μη ε. Έχουμε και τοπικά μη μη αλλά από πρακτικής πλευράς δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη αποστολή για αυτά τα ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο ασχολούνται για την ιστορία, για την ταυτότητα των κρατών. Αλλά εμείς δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε την ευρωπαϊκή σαγένεια με την εθνικότητα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία με τα τοπικά ΜΜΕ. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή να βρεθεί ο χώρος. Δεύτερο, νέα μέσα επικοινωνίας, τα κοινωνικά δίκτυα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα λείπει η Ευρώπη. Σε εκατοντάδες ιστοσελίδες που συμβουλεύονται εκατομμύρια πολιτών. Ασχοληθήκαμε εμείς για τη νέα μορφή αναμετάδοσης περιεχομένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ας πούμε, τα σχολεία χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μέσα μέσω διαδικτύου. Θα έπρεπε να δοθεί προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα των νέων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων. Και με τον συνάδελφο Μιγάσκι, εμείς βιώσαμε στην Πολωνία αυτή την τραγωδία τώρα τελευταία. Όλη η πολωνική κοινωνία, τα ΜΜΕ αναρωτήθηκαν, μα σε τι στοχεύει η δημόσια σφαίρα, κβο η Πολωνία, κβο η Ευρώπη, πού πηγαίνουν λοιπόν. Ντόμινε. Πρέπει να αναθέσουμε περισσότερες ευθύνες στα ΜΜΕ αντί μόνο να τρέχουμε σε βοήθειά τους όταν μας χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για μία σύντομη παρατήρηση στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πακ. Από τη δικιά μας ε, πλευρά χαιρετίζουμε την έκθεση του κυρίου Λόκεγκαρντ, ο οποίος αναφέρεται σε ένα ενδιαφέρον θέμα, δηλαδή πώς θα βελτιώσουμε την επικοινωνία ε, για το τι κάνουμε όλοι εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Η ανάλυση του της παρούσης κατάστασης είναι πολύ ορθή. Απέχουμε πολύ από το ευρωπαϊκό πρότυπο. Οι επικοινωνίες γίνονται στο εθνικό επίπεδο επικοινωνίας και ε, δεν ε, τα δημόσια θέματα δεν έρχονται ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη, ούτε τέταρτη θέση. Όσον αφορά τα μέσα, ε, ναι, ε, υπάρχουν νέα μέσα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν και θέλουμε ε, να εργαστούμε καλύτερα με τον τύπο. Εάν εξετάζω τις τρεις προτάσεις, τη βαθμολόγηση για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, και νομίζω ήταν περισσότερο για την τηλεόραση, από πλευρά μας δεν ε, έχουμε κάνει όπως ζητήθηκε μία ποιοτική αξιολόγηση των ε, τηλεοπτικών προγραμμάτων. Έχει γίνει ποσοτική, δηλαδή πώς η Ευρώπη υπάρχει εβδομαδιαία, ημερήσια, μηνιαία ε, στην τηλεόραση. Και μπορούμε να σας πούμε ότι αν θέλετε τέτοιες προφορίες μπορούμε να σας τις παράσχουμε. Βεβαίως, εμείς ε, δεν μπορούμε να σας δώσουμε τη βαθμολόγηση, αλλά μπορούμε να σας δώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Όσον αφορά τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ε, βεβαίως συμφωνούμε με ορισμένα από αυτά που είπατε όσον αφορά την ανεξαρτησία ε, αλλά ένα, μια κυβέρνηση, ένα κράτος ε, δεν πρέπει να παρακολουθεί μόνο τι γίνεται πολιτικά εθνικά αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχουμε καμία δυσκολία με αυτό και υπάρχει ένας αριθμός κρατών που ήδη έχουν παρεμφερεί μέτρα και θα ήθελα να τα αναφέρω, διότι θα σας αναφέρω τώρα μία φράση της γαλλικής νομοθεσίας για τη δημόσια τηλεόραση στη Γαλλία ότι η France Television πρέπει να εντάξει την ευρωπαϊκή διάσταση στα προγράμματα κτλ. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο άρθρο ή στην νομοθεσία που αφορά την, τη ε, δημόσια τηλεόραση όχι επί της ουσίας αλλά ότι θα πρέπει να αναφέρονται σε ευρωπαϊκά θέματα ή ε, την δημόσια τηλεόραση τηλεόραση. Οπότε εμείς συμφωνούμε με τα στοιχεία που αναφέρει ο κύριος για στην έκθεσή του. Επίσης, ε, το ε, καθήκον ε, οι ανταποκριτές να παρακολουθούν τι γίνεται εδώ και στο Στρασβούργο νομίζω ότι πολύ σωστά δεν θα συμφωνούσαμε γιατί θα ήμασταν σε άμεσο ανταγωνισμό με αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν και ε, ε, έχουμε διαφορετικό γραπτό τύπο ε, εδώ. Όντως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση για την Ευρώπη η ε, τα σχολεία αλλά επειδή μας προέτρεψε η Πρόεδρος να μην ξεπερνάμε το ε, μικρό χώρο θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ για όλες τις επεμβάσεις. Ο κύριος Λόκεργαρντ έκανε μία έκθεση η οποία προκάλεσε πολύ επικοδομητική κριτική εγώ νόμιζα ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα του. Αυτό θα ήταν καλύτερο αντί ε, να ασχοληθεί με όλα διότι μιλάμε για δημοσιογραφία και νέα μέσα ενημέρωσης οπότε ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθεί καλύτερο ε, σε ε, αυτά τα δύο θέματα και συμφωνώ με τα υπόλοιπα αλλά κατά τα άλλα αναφέρθηκαν πολλά θέματα που είναι σημαντικά και πρέπει να σας πω ότι το 14 δεν έχει καμία θέση εδώ όπου αναφέρεται η ε, κριτική αξιολόγηση που δεν έχει καμία, καμία θέση στο θέμα μας άρα θα έπρεπε να διαγραφεί. Και μήπως την έκθεση, όπως είπε, ελέγχθηκε εδώ σήμερα, στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, ε, ε, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να προωθηθούν, δηλαδή ε, πλατφόρμες του διαδικτύου και εάν προωθήσουμε αυτές τις ε, ε, πρωτοβουλίες ήταν πολύ πιο επιτυχής η έκθεσή σας. Δεν μπορούμε πλέον να συζητήσουμε, θέλετε να απαντήσετε κύριε Λόκερ, αλλά σύντομα γιατί δεν έχουμε πια πολύ χρόνο. Ναι, φυσικά και θα είμαι πολύ σύντομος, διότι αλλιώς θα ξεκινούσα μεγάλο διότι έχω να ξεκινήσω μεγάλο ταξίδι. Άκουσα πολύ καλέ ε, παρεμβάσει από όλου και αυτό το περίμενα, διότι είναι θέμα που απασχολεί του περισσότερου από, από εμά. Πολύ σύντομα θα ήθελα να, τονίσω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι το είπα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου, αλλά θα το ξαναπώ. Είμαι και εγώ δημοσιογράφο. Επί 30 χρόνια ήμουν. Ε, δεν θα μπορούσα ποτέ να, να σκεφτώ καν να ε, παραβιάσω την ε, ελευθερία, την ανεξαρτησία του δημοσιογράφου. Κάποιες ε, προτάσεις, ναι, ίσως ξεπερνούν λίγο τα όρια, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι με κανέναν τρόπο δεν θα παραβιάσουμε το δικαίωμα αυτό. Από την άλλη θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, αντιδράμε αυτόματα σε πολλά από τα πράγματα που εδώ. Έχουμε 40 χρόνια ε, και υπάρχει σημαντική απουσία προτάσεων για το πώς θα προχωρήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πω σε όλους ότι αν όλοι είσαστε διατεθειμένοι να ε, ξεκινήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό με το σωστό πνεύμα, τότε θα είμαι και εγώ απόλυτα ανοιχτό όσον αφορά τη διατύπωση των διαφόρων θεμάτων. Απλά θα ήθελα να τονίσω ε, όπως υπόθηκε από διάφορους, δεν πρόκειται για προσβολή των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. Και εγώ δημοσιογράφος είμαι. Ε, το θέμα είναι κάποιοι από εμά να μπούμε στο σύστημα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι καινοτόμο. Από την άλλη, είναι μια νέα ιδέα και θα πρέπει να σκεφτούμε καινοτόμα, διότι αλλιώ θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί που είμαστε τώρα, δηλαδή στο πουθενά. Προσλέπω λοιπόν στι ε, καλέ διαπραγματεύσει και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε ε, σε ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο επιτέλους να οδηγήσει σε κάτι συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λόκεργαρτ. Ε, μπορούμε τις προτάσεις μας να τις υποβάλουμε γραπτός μέχρι την 4η Μαΐου. Παρακαλώ να παρουσιάσετε τροπολογίες για να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση την οποία, η οποία έχει διαγραφεί και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Λόκεργαρτ θα παρουσιάσει τροπολογίες. Ευχαριστώ όλους γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον, σε αυτή η συζήτηση αλλά όταν έχουμε εμπειρογνώμονες δεν έχουμε πλέον επαρκή χρόνο και μετά τρέχουμε. Ε, πολύ σωστά κάνατε αυτό διότι ότι το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε με τον Ιβο Μπέλετ και επειδή είμαι πάντοτε γενναιόδορη υποκύπτω αλλά ελπίζω ότι οι επόμενοι ομιλητές θα είναι σύντομοι. Ερχόμαστε τώρα στο το θέμα της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στην ψηφιακή εποχή, το μέλλον του διτού συστήματος, εισηγητής ο κύριος Μπέλετ και έχει καλέσει και δύο ανεξάρτητους εισηγητές, μία ε, εκπρόσωπο από την Ρουμανία και ε, το έγγραφο θα προχωρήσει και θα υποβληθεί τον Ιούνιο. Δεν έχουμε προχωρήσει δηλαδή τόσο πολύ όσο και με τον κύριο Λόκεγκαν. Ε, στις 22 Ιουνίου θα συζητήσουμε το σχέδιο της εκθέσεως και το Σεπτέμβριο πλέον θα ψηφίσουμε, δηλαδή το Σεπτέμβριο θα τελειώσει η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ε, έχουμε ε, καθυστερήσει λίγο τον κύριο Μαρτίνες ο οποίος θα έρθει σε 45 λεπτά αντί για σε μισή ώρα οπότε έχουμε 45 λεπτά και παρακαλώ να μην ε, ξεπεράστε το χρόνο αυτό διότι δεν θα μπορέσω πλέον να επιτρέψω εξαιρετικούς εισηγητές και παρόλο που αυτό βοηθά τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ντόρι, θα είμαι πολύ σύντομος διότι όπως είπε, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα αναφερθώ στην εμβέλεια της εκθέσεως αυτής και στα βασικά θέματα διότι αναφερόμαστε εις ε, τη δημόσια ε, ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία πώς λειτουργεί στην ψηφιακή εποχή και το διτό σύστημα. Αυτά είναι τα ουσιαστικά στοιχεία. Όταν μιλάμε για διτό σύστημα, μεικτό σύστημα δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών στα μέσα ενημέρωσης που εξασφαλίζουν την πολυμορφία και την ποικιλομορφία όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο του Άμστερνταμ που είναι πολύ σημαντικό σε σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς όμως ε, υπάρχει το πρόβλημα ότι το τοπίο της ε, ε, ραδιοτηλεόρασης ή στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ακόμη και υπαρξιακά και εδώ αναφερόμαστε στην έλλειψη σωστής διακυβέρνησης προσβάσεως σε νέες ψηφιακές πλατφόρμες και σε έλλειψη ανεξάρτητης χρηματοδότησης πράγμα το οποίο πλήττει διάφορα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα σημείο όπου πολλοί από τους ε, ραδιοτηλεοπτικούς ε, υπευθύνου ε, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να, να αντισταθούμε στην υπερβολική αντιμετώπιση και θα πρέπει να ε, αναφερθούμε εις ε, την ε, έλλειψη αυτή με διαφορετικό τρόπο από αυτό που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης διότι όταν μιλάμε για ανεξαρτησία των, των δημοσίων σταθμών όταν μιλάμε ε, για ανεξάρτητους κανόνες ε, για αυτά τα είδη των ε, ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε διάφορους κανόνες. Άρα αυτό είναι το, η πιο βασική μας πρόκληση δηλαδή όσον αφορά ε, το μέλλον αυτών των υπηρεσιών και αναφερόμαστε και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Σε αυτή λοιπόν την, ε, ε, σε αυτό το περιβάλλον με διάφορες πλατφόρμες υπάρχει δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός μεταξύ των των διαφόρων ε, μέσων ενημέρωσης παρά μόνο με τις εφημερίδες και οι εκδότες των εφημερίδων και των περιοδικών προσπαθούν να τοποθετηθούν στο διαδίκτυο και έχουν μειώσει σημαντικά τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία έτη το εισόδημά τους χρειάζονται εισόδημα δηλαδή ε, θα έπρεπε τα περιοδικά και εφημερίδες να έχουν επιπρόσθετο εισόδημα από το ίντερνετ αλλά το Google παίρνει 50% της αγοράς διαφήμισης ε, και οι εκδότες δεν μπορούν να αντιταχθούν ε, στην, ε, στο ελεύθερο διαδίκτυο, το δωρεάν διαδίκτυο στο οποίο έχουν πρόβληση, έχουν πρόσβαση τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και βλέπουμε ότι τώρα δεν χρειάζεται μόνο να αναφέρεται κανείς ε, στην, ε, στα παραδοσιακά μέτρα μέσα αλλά επίσης και σε αυτά που έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και βεβαίως κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και γι' αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρτισε ε, επί του θέματος ε, μία ανακοίνωση ε, για την ραδιοτηλεόραση και στο 2009 που λέγει ότι θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιοι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες οι οποίες όταν προσφέρουν νέες υπηρεσίες στο διαδίκτυο θα πρέπει ε, ε, ε, καταρχήν να έχουν αξιολογηθεί. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μία διάταξη η οποία θα αναφέρεται σε διαβούλευση δημόσια προτού εφαρμοστεί. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι λέγουν ότι η ε, δημόσιες αυτές υπηρεσίες θα έπρεπε ε, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή ε, στο διαδίκτυο και από την άλλη πλευρά οι υπηρεσίες αυτές λέγουν ότι δεν θέλουν να περιοριστούν στις δραστηριότητες τους για το διαδίκτυο στην ψηφιακή εποχή. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε νέα πρότυπα, να μπορέσουν να συνεπάρξουν όλα αυτά τα συστήματα στο διαδίκτυο και βεβαίως επ' αυτού θα ήθελα να έχω πολλές προτάσεις από εσάς κατά τη συζήτηση, όχι μόνο για να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά για να διατυπώσουμε νέα πρότυπα. Δεν σκοπεύω εδώ να ε, υπησέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά θα αναφέρω ορισμένες ιδέες μου. Ε, καταρχήν να να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου των μέσων και ε, στο διαδίκτυο και των εφημερίδων και του τύπου δηλαδή ε, να υπάρχει ε, μια συνεργασία. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, για το Google, για διάφορες άλλες υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Θα μπορούσαν ε, να δημιουργήσουμε ε, διάφορα μέσα με τα οποία το Google, παραδείγματο χάρη, θα υποχρεωθεί να συμβάλλει στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να υπάρξουν ελάχιστα κριτήρια για την είναι διακυβέρνηση στο διαδίκτυο και ε, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ και πολλά θέματα. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμά μου. Το διτό σύστημα κατά τη γνώμη μας δεν είναι κάτι στατικό, είναι μία πρόοδος στις εργασίες μας και προσβλέπουμε σε μία υγιή ε, ισορροπία μεταξύ ε, του γραπτού τύπου και ε, ε, των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στο διαδίκτυο και εμείς θα προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό πρότυπο κατά τρόπον ώστε ε, να ε, αναγνωρίσουμε ότι πολλά, πολλοί συμμετέχοντες σε αυτό το σύστημα περνούν πολύ δύσκολες μέρες και ελπίζω ότι με την ανταλλαγή απόψεών μας και η δικιά σας ε, συμμετοχή θα επιτρέψει ένα βιώσιμο αηφόρο μέτρο διότι και αυτά αναφέρονται στην ελευθερία και στη δημοκρατία. Τώρα δίνω το λόγο για πέντε λεπτά, χωρίς να έχουμε και πολύ χρόνο, στην κυρία Αβαντίνη, η οποία είναι υπεύθυνη στη Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εθνική οπτική και να γίνω πιο συγκεκριμένη όσον αφορά τη βασική δομή που παρουσίασε ο κύριος Μπέλετ. Στη Ρουμανία ο Πρωθυπουργό σε μια υπόθεση ζήτησε ε, να έχει κάθε βδομάδα 30 λεπτά δικά του στην τηλεόραση. Δεν είναι φανατικός κομμουνιστής, δεν είναι δεινόσαυρος, ε, διδάσκει συνταγματικό δίκαιο. Ξέρει λοιπόν τα πράγματα αυτά, ωστόσο συνεχίζει να ζητά το χρόνο του, μάλλον όχι για τον ίδιο αλλά για την κυβέρνηση. Η ιδέα είναι στο μυαλό όλων η δημόσια τηλεόραση να εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Και το παράδειγμα αυτό δείχνει το βασικό πρόβλημα των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στα νέα κράτη-μέλη. Ε, έχουν ένα πρόβλημα ταυτότητας. Εξυπηρετούν το κοινό, το κράτος, Άλλωστε είναι εθνικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έδειξε ότι μόνο το 20% των ε, ραδιοφωνικών καναλιών και το 30% των τηλεοπτικών, και μιλάμε για εκατοντάδες κανάλια, έχουν πολιτιστικά προγράμματα. Όλα τα άλλα είναι βασικά ψυχαγωγία, και πότε πότε ειδήσει. Από τη μία λοιπόν έχουμε κατάχρηση μιας υπηρεσίας, έχουμε μια υπηρεσία υποπίεση από την κυβέρνηση, από την άλλη έχουμε σημαντική ανάγκη για τις υπηρεσίες αυτές. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, στην κορυφή, βρίσκονται τα δημόσια κανάλια όσον αφορά την, ε, τις πολιτιστικές εκπομπές. Έχουμε προβλήματα διακυβέρνησης, ναι, διότι δεν ξέρουμε ποιος ουσιαστικά διευθύνει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έχουμε προγράμματα χρηματοδότησης και να σας αναφέρω μια άλλη ιστορία. Δημοσιογράφος, είμαι ιστορίες λέω. Το 2005 ο πρώην Διευθυντής της Δημόσιας ε, Τηλεόρασης απολύθηκε λόγω ε, διαχειριστικών ε, θεμάτων, αλλά σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Δύο χρόνια αργότερα ο διάδοχος του αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη θέση του λόγω των ε, σημαντικών δαπανών και της τρύπας στον προϋπολογισμό. Αλλά η δημόσια τηλεόραση ήταν πολύ δημοφιλής τότε. Τι θέλουμε εμείς από τις υπηρεσίες αυτές. Θέλουμε οικονομική απόδοση. Τι είδους υπηρεσία θέλουμε. Η κατάσταση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά τη Ρουμανία. Για παράδειγμα, στη Σλοβακία 14 διευθυντές σε 18 χρόνια είχαν και η Ουγγαρία επί δύο χρόνια προσπαθεί να βρει πρόεδρο για τις δημοσίες αυτές υπηρεσίες. Είναι σαφές λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση. Τα τελευταία 18-20 χρόνια η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαριστεί. Γνωρίζω καλά το θέμα της επικουρικότητας. Γνωρίζω καλά τις πτυχές που αφορούν τον ανταγωνισμό που ανέφερε ο κύριος Πέλετ. Ωστόσο, Πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για κάποιο είδους δομές ώστε οι δημόσιες ραδιοτηλεφωνικές, ε, ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες να μπορούν να αναπτυχθούν στη νέα αυτή εποχή. Εγώ θα ήθελα να δώσω διαφορετική έμφαση από τον, έμφαση από τον κύριο Μπέλετ, να μιλάμε για δημόσιες ε, ραδιοτηλεοπτικέ υπηρεσίες και τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μας οδηγήσουν ακριβώς εκεί. Εάν σκεφτόμαστε του τους θεσμούς, φορεί, τους φορείς, ίσως να έχουμε ήδη χάσει το παιχνίδι. Εγώ θα σας καλούσα να σκεφτούμε το κοινό, τους ακροατές, τους θεατές, τους καταναλωτές των υπηρεσιών αυτών. Στην προηγούμενη, στα πλαίσια της προηγούμενης έκθεσης ε, ακούσαμε πληροφορίες για την νεολαία. Ξέρουμε από πού παίρνει η νεολαία τις πληροφορίες της. Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Και αν αναλύσουμε την αγορά, όσα έχει αυτή τη στιγμή, και πάλι θα έχουμε χάσει το τρένο. Εάν η καλή νεράιδα μπορούσε να μου εκπληρώσει μία ευχή, εγώ θα ήθελα μελέτη σχετικά με το πώς συλλέγουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες τα παιδιά, ηλικίες 9 με 12 και 12 με 15. Έτσι θα έχουμε το περιφέρειο να κατανοήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για να έχουν τα παιδιά αυτά πρόσβαση σε ε, δημόσιες υπηρεσίε. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εκπομπές, μιλάω και για νέε πλατφόρμες, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Νομίζω ότι 15 χρόνια από σήμερα το περιβάλλον των μέσων μαζική ενημέρωση θα είναι τελείως διαφορετικό από, από ό,τι είναι σήμερα. Και εάν προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε μόνο αυτά που έχουμε τώρα, θα έχουμε χάσει το τρένο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά, το έγγραφο έχει διανεμηθεί αγγλικά και συνοψίζει αυτά τα οποία θα πω σήμερα. Ο κύριος Κολέτα με, Μπελέτ με βοήθησε πολύ με την εισαγωγή του διότι υπενθύμησε ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης που αλλάζει όλες τις παραμέτρους των μέσων ενημέρωσης και υποχρεώνει και τα δημόσια και τα ιδιωτικά μέσα να ξανασκεφτούν ε, το τι μέλη γενέστε με τις οργανώσεις τους και την κατανομή των πόρων. Γενικά, ε, όσον αφορά τα ε, ψηφιακά μέσα, το σύστημα είναι νέο και δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη. Δεν μπορούμε δηλαδή σήμερα ε, έναντι αυτής της κατάστασης ασταθίας, να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν όπως ε, έχει γίνει στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης των δημοσίων μέσων. Αυτό το οποίο πρέπει να υπενθυμίζουμε είναι η ελευθερία εκφράσεως που δεν θα υπάρχει χωρίς οικονομική ανεξαρτησία των ιδιωτικών μέσων. Γι' αυτό και ε, πρέπει ε, εις ε, το ψηφιακό τομέα να υπάρχουν βιώσιμα επιχειρησιακά πρότυπα για να μπορούν να αξιοποιηθούν τα περιεχόμενα τα οποία έχουν εκπονηθεί χωρίς η αξία αυτή να καταστραφεί από αθέμητο ανταγωνισμό. Το θέμα που τίθεται, όπως είπε ο κύριος Μπουλέτ, διαφέρει αναλόγως των κρατών μελών, διότι τα δημόσια μέσα δεν αναφέρονται στο ίδιο σημείο και ε, υπάρχουν ορισμένες πιο πλούσιες χώρες όσον αφορά την προσφορά ε, μέσων που έχουν, αλλά θα ήθελα να την προσοχή σε μικρές χώρες όπως το που υπό, υφίστανται την πίεση ε, των γειτονικών χωρών και των εκπομπών των μέσων τους και όπου προκύπτουν ορισμένες δυσκολίες που ίσως δεν αντικατοπτρίζονται στα μεγάλα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τρεις άξονες ουσιαστικά. Καταρχήν, διαπιστώνουμε ότι είναι δύσκολο να καταρτιστούν νέα πρότυπα οικονομικά στο ψηφιακό σύστημα. Το δεύτερο και αυτό είναι απολύτως νόμιμο ε, ε, είναι να γνωρίζουμε τι πρέπει να είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση το 2010 και ακόμη περισσότερο στο μέλλον και τρίτον να επινοήσουμε δημιουργικά μία εναρμόνιση του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε αυτό το χώρο. Άρα, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για τη δυσκολία κατάρτισης οικονομικών μοντέλων, θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε διάφορα θέματα, ε, δηλαδή ε, να, το, το ακουστικό τώρα να γίνει μια σταθερή εικόνα στο διαδίκτυο πράγμα το οποίο είναι κάτι νέο και δημιουργεί ε, μια μεγάλη, ένα μεγάλο ανταγωνισμό. Δεύτερον, υπήρχε ε, το ίντερνετ ε, ένας κατακαιρματισμός της διαφήμισης που ξεχώριζε το οπτικοακουστικό από τα θεσμικά θέματα και από τα θέματα των αυτοκινήτων και άλλες διαφημίσεις. Ενώ τώρα όλα μπορούν να στηρίζονται στο ψηφιακό σύστημα. Και αυτού του είδους η διαφήμιση είναι με τοπικά αντίθετη από την διαφήμιση στον τύπο. Αυτό λοιπόν εντείνει τον ανταγωνισμό. Υπάρχει και ένας δεύτερος με δεύτερο επίπεδο με τοπικού ανταγωνισμού λοιπόν. Έχουμε επίσης το πρόγραμμα των νέων operators, νέων λειτουργών, που είναι, που είναι οι οργανισμοί τηλεφωνίας που οργανώνονται καθέτος, ε, ε, υπάρχουν ε, όλα, όλοι οι μηχανισμοί αναζήτησης που καρπούνται των εργασιών του τύπου. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς αυτά να τα αγνοήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε τα διάφορα επίπεδα εξουσίας, από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι το ευρωπαϊκό επίπεδο, να κοιτάξουν, να ρυθμίσουν την αγορά για να διασφαλίσουν τον πλουραλισμό, το περιεχόμενο και την προστασία επίσης των δημιουργών. Και η αλυσίδα των αξιών να βρει τη θέση της όλοι όσοι παράγουν και δημιουργούν θα πρέπει να ανταμείβονται. Το δημόσιο χρήμα δεν θα πρέπει να χρησιμεύει στην στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή. Το είπα και προηγουμένως. ότι υπάρχει στρέβλωση στον τομέα της διαφήμισης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν στα, ότι τα δημόσια ΜΜΕ σίγουρα πρέπει να βρίσκονται στο ίντερνετ, αλλά πρέπει να βρίσκονται στο ίντερνετ ούτω ώστε η παρουσία τους να εγγυάται την αξία τους και το ρόλο τους και την αποστολή τους. Δηλαδή, σήμερα θα πρέπει να να αναρωτηθούμε ποια είναι η αξία αυτής της νέας υπηρεσίας των δημοσίων ΜΜΕ στον ίντερνετ. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει δημόσια χρηματοδότηση για την εκπλήρωση του ρόλου των ΜΜΕ όταν υπάρχει λοιπόν ρόλος δημοσίου ωφέλους και κοινού ωφέλους, τότε θα πρέπει να δοθεί χρηματοδότηση. Εάν το κοινό έχει πρόσβαση πλουραλιστικά και διαφοροποιημένα στην πληροφόρηση, θα πρέπει κανείς να αναρωτηθεί γιατί θα πρέπει να δώσουμε δημόσια κονδύλια σε οικονομίες οι οποίες πλήττονται από παντού, για να κάνουν τα δημόσια ΜΜΕ την ίδια δουλειά των ιδιωτικών. Και αυτή είναι μια δραματική τάση, την παρατηρούμε από το 80 και μετά. Δηλαδή βλέπουμε τον δημόσιο τομέα να τρέχει πίσω από τα, από τα ιδιωτικά μέντια σε έναν ανταγωνισμό απόλυτα άγωνο και αντιπαραγωγικό. Ας πούμε αυτό γίνεται με τα αθλητικά δικαιώματα. Η κυρία Πάκ εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά λέει με μικρόφωνο η κυρία Πακ. Και δίνουμε το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους και στην Κομισιόν. Ο κύριος Δράτσεμπράι από την Κομισιόν. Χωρίς μικρόφωνο Κομισιόν. Με μικρόφωνο Κομισιόν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτή την συζήτηση η οποία είναι επίκαιρη και σημαντική. Δηλαδή, ε, τι αλλάζει το τοπίο στην ε, ευρωπαϊκή ραδιοτηλεόραση. Ε, υπάρχουν και δημόσιοι και ιδιωτικοί δημόσιες και ιδιωτικές εκπομπές και πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, την ανεξαρτησία της και την πρόσβαση σε διάφορες πλατφόρμες. Ε, στο διαδίκτυο διότι λέχθη ότι σύμφωνα με την ε, μέθοδο που με την ανακοίνωση που υιοθέτησε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντούμε ε, σε πολλά από αυτά τα θέματα και το πιο εύκολο είναι η πρόσβαση στις πλατφόρμες διότι υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο σχετικά με τη διαφοροποίηση των εκπομπών δημοσίου συμφέροντος όπου ε, λέγεται ότι θα υπάρχει πρόσβαση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή αυτή είναι η απάντηση στην αίτηση την οποία είχε κάνει η ΕΜΠΑ ε, και αναφέρεται αυτό που ελέγχθη στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και να αξιολογήσετε τις στρεβλώσεις της αγοράς που θα δημιουργούσε η προσφορά του δημοσίου ε, ε, για τα δημόσια μέσα. Και βεβαίως ε, υπάρχουν ορισμένες αιτιολογισμένες στρεβλώσεις όσον αφορά όμως την ανεξαρτησία θα ήθελα και πάλι να παραπέμψω στην ανακοίνωση η οποία συνδέει το πρώτο θέμα με αυτό. Δηλαδή, η ανακοίνωση εξηγώντα το τι υπάρχει στη συνθήκη και στο πρωτόκολλο του Άμστερνταμ αναφέρει ότι δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει ποια προγράμματα θα προσφέρονται και θα χρηματοδοτούνται από πλευράς γενικού συμφέροντος ή να αμφισβητήσει τη φύση ορισμένων από αυτά τα προϊόντα είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτός. Απλούστατα η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει τα προφανή λάθη. Και τέλος αναφέρομαι στο θέμα της σωστής διακυβέρνησης. Και ίσως θυμάστε τη συζήτηση την οποία είχαμε όταν ε, συζητήσαμε για την οδηγία για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης ε, που η θέση των κρατών ε, μελών ε, είχε επίσης εξεταστεί και αυτό δεν αναφέρεται μόνο εις την διακυβέρνηση των μέσων των δημοσίων μέσων εκπομπής προγραμμάτων αλλά ε, σε όλα τα σημεία τα οποία ενδέχεται να δυσχεραίνουν εδώ τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ε, η κυρία Κάμα Εύατ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μετά τον εκπρόσωπο της Κομισιόν μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Είχα μια συνάντηση πριν με τον Ιβο Πέλετ και μαζί σκεφτήκαμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάει η έκθεση αυτή. Και πιστεύω ότι πολύ σημαντικό και αποφασιστική σημασία είναι ότι θα πρέπει να εργαστούμε με βάση το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ και της ε, ανακοίνωσης ε, για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα Τη περσινή χρονιά, διότι εκεί ήδη έχουν ληφθεί βασικές θεμελιώδει αποφάσεις. Στην ε, Γερμανία έχουμε τώρα τη διαφωνία σχετικά με το τεστ των τριών επιπέδων και στη συζήτηση αυτή που γίνεται στη Γερμανία αυτή τη στιγμή φαίνεται πόσο ε, αποτελεσματικό είναι αυτό, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο συμβιβασμός ε, που βασίζεται στα, στις αποφάσεις της Κομισιόν. Εάν αυτό αποτελέσει τη βάση για τις ε, περαιτέρω αποφάσεις μας και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό στην Επιτροπή μας, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια καλή έκθεση στραμμένη προς το μέλλον. Αυτή είναι όπως προϋπόθεσή μου, θα πρέπει αυτή να είναι η βάση για τις περαιτέρω εργασίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πολύ να αναφέρω ότι η πρωτοβουλία για την έκθεση αυτή προέκυψε από τα προβλήματα που έχουμε κυρίως στα νέα κράτη-μέλη που ε, προσχώρησαν ε, το 2004, ε, καθώς και προβλήματα που υπάρχουν σε, κάποιες, σε κάποια παλιά κράτη-μέλη, το γεγονός δηλαδή ότι όταν λέμε δημόσια ε, ε, ραδιοτηλεόραση στα διάφορα κράτη-μέλη δεν εννοούμε τα ίδια πράγματα και το παράδειγμα που ακούσαμε από τη Ρουμανία το δείχνει αυτό. Σε πολλά δυτικά κράτη-μέλη έχουμε την κρατική τηλεόραση. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ισορροπία ανάμεσα ε, στην ε, τηλεόραση δημοσίου δικαίου που έχει συγκεκριμένη υποχρέωση όσον αφορά την εκπαίδευση, την κουλτούρα. Από την άλλη έχουμε την ιδιωτική ε, ραδιοτηλεόραση που φυσικά υπόκειται στους σχετικούς νόμους αλλά, που, αλλά όπου θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει σκοπό να βρει ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και την ιδιωτική. και να βοηθήσει την κάθε μία από αυτές για να κάνει τη δουλειά τους. Πολύ σωστά αναφέρθηκε το πρόβλημα του ανταγωνισμού. Έχουμε κανάλια τα οποία χρηματοδοτούνται με χρήματα των φορολογουμένων ε, που ανταγωνίζονται άλλα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι θέμα το οποίο, ε, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Η κυρία Καμερέβερτ ε, ανέφερε το πρόβλημα αυτό. Πιστεύω ότι γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που προκύπτουν από το πρόβλημα αυτό ο Ιβο Μπέλετ ανέφερε την πολύ καλή δουλειά του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει κάνει πολύ προπαρασκευαστική εργασία. Δεν χρειάζεται να ξαναφεύγουμε τον, τροφό, τον τροχό, συγγνώμη, μπορούμε να βασιστούμε στη δουλειά αυτή. Θα παρακαλούσα τους συναδέρφους να να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Είπαμε στον κύριο Μαρτίνε να έρθει αργότερα, αλλά τώρα τελειώσαμε νωρίτερα. Υπάρχει άλλο που να θέλει να πάρει τα λόγο. Αν όχι, να δώσω το λόγο στον Ήβο. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω στα Ολλανδικά, κυρία Πρόεδρε. Αυτό το οποίο είπατε είναι ουσιαστικότατο. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία, τη συνύπαρξη Αυτό γράφτηκε και στην περσινή ανακοίνωση για τα ραδιοτηλεοπτικά. Πώς να τα διαχειριστούμε όμως όλα αυτά. Δηλαδή από τη μανιά τα δημόσια ΜΜΕ και από την άλλη τα ιδιωτικά. Και μετά φυσικά ανταγωνισμός μεταξύ των δύο και του τύπου. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια καλή ισορροπία. Όλα αυτά είναι σημαντικότατα για τη διασφάλιση του πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Πρέπει να αποφύγουμε να περιορί... τον περιορισμό της δυναμικής των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών μέσων στο ίντερνετ. Θα πρέπει και αυτά να έχουν τον επαρκή τους χώρο στο ίντερνετ για να κάνουν τη δουλειά τους. Ξαναλέω λοιπόν, αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ όλων. Δεύτερο, δεν πρέπει να πέσουμε σε μία στήρα συζήτηση. Μιλήσατε για τα νέα κράτη-μέλη, αλλά δέστε και τα παλιά κράτη-μέλη τι γίνεται. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε εμείς και να λέμε ορίστε η Ιταλία, η Γαλλία, ή το Βέλγιο ή δεν ξέρω τι. Πρέπει να έχουμε αρχές και όχι να φορτώνουμε λάθη στους νέους. Ε, ε, πρέπει να έχουμε ιδέες λοιπόν ακούσαμε πυρογνώμονε σήμερα. Πρέπει να ακούσουμε όμως και άλλους για να ολοκληρώσουμε την άποψή μας για να έχουμε και φρέσκο και καινοτόμο υλικό για τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χρόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο για την ψηφοφορία. Έχουμε λοιπόν το χρόνο πριν το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο θα ψηφίσουμε οριστικά. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Για τους συναδέλφους που δεν είναι παρόντες, έχουμε το εξής πρόβλημα. Θα έχουμε μάλλον πάλι Κάουζα Ιτάλια. Παρακαλώ την έκθεση αυτή να την δούμε ως μια γενική αντικειμενική έκθεση χωρίς να κατηγορούμε την Ιταλία, τη Ρουμανία ή δεν ξέρω ποιον, διότι έτσι θα καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων. Θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το θέμα χωρί να αναφέρουμε ονόματα, διότι αυτό δεν φέρνει τίποτα. Δεν είναι έκθεση που αφορά τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωση. Έχει να κάνει με το διτό σύστημα, την ε, δημόσια και την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση και είναι πολύ πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά και σοβαρά. Παρακαλώ του συναδέρφους που πάντα θέλουν να, ε, να ενσωματώσουν τα θέματα αυτά σε κάθε έκθεση, παρακαλώ να μην το κάνουν. Δεν είναι αυτός ο κατάλληλος χώρος να αρχίσουμε πάλι να αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα. Δεν βοηθάει αυτό το αντικείμενό μας. Δεν θέλω να εξοραίσω τα πράγματα. Έχω το ίδιο πρόβλημα που έχετε όλοι σας με το πρόβλημα αυτό, αλλά θα ήθελα να περιοριστούμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα, το διτό σύστημα δηλαδή, πώς μπορούμε να τα ρυθμίσουμε αυτά και πώς μπορούμε στο νέο ψηφιακό κόσμο να πετύχουμε ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης στον τομέα του ίντερνετ. Άλλωστε και στην ανακοίνωση της Κομισιόν ε, περιοριζόμαστε στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρωθυπουργό, θα μπορούσα σας είχα αφήσει να μιλήσετε περισσότερο, λυπάμαι δεν το ήξερα νωρίτερα. Ε, ως πρόεδρος πρέπει να φροντίζω να επιβάλλω την τάξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι τώρα στο θέμα 12 της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις στις αποφάσεις των συντονιστών ε, της χθεσινής συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση... Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών και ε, φτάνει ο συνάδελφος Μαρτίνες. Παρακαλώ να παραμείνετε εδώ για να ακούσουμε τι έχει να μας πει σχετικά με το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, που είναι πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Παλιαδέλη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ίσως θα ε, μου επιτρέψετε να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής μας. Να σας θυμίσω ότι προσπαθήσαμε να, τα, να εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα του βραβείου Λουξ στα διάφορα κράτη-μέλη. Έκανα ό,τι μπορούσα. Το, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στις 9 Μαΐου στη χώρα μου και στη Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα γίνει ε, δημόσια δωρεάν προβολή για το κοινό της ε, ταινία ε, που κέρδισε και θα γίνει και συζήτηση σχετικά με αυτήν. Ελπίζω του χρόνου να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και να μπορέσουμε να το επιδείξουμε αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να συνεχίσω. Εγώ το έκανα με την συνάδελφο την κυρία Ράνα στο, ε, στο Γκράτς. Ε, είχαμε ελεύθερη είσοδο στο σινεμά και έγινε και συζήτηση και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και να σας δώσω ε, και μια πληροφορία. Όλοι οι δημόσιοι ευρωπαϊκοί χώροι, δηλαδή οι αντιπροσωπείες στα διάφορα κράτη-μέλη, έχουν υποσχεθεί ότι κατά διάρκεια τη Ευρωπαϊκή Εβδομάδας θα δώσουν τη δυνατότητα προβολής τη ταινία αυτή. Γίνεται λοιπόν όλο και πιο ορατή. Σα ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωσή σας αυτή και σα ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Λοιπόν, αγαπητέ Μίγκελ Άγγελ Μαρτίνες Μαρτίνες. Είσαι παλιός φίλος από τις ε, μέρες που ήμασταν μαζί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Χαίρομαι πολύ που ήρθες για να μας παρουσιάσει στο σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στο θέμα για να συζητήσουμε μετά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ντόρις. Πράγματι. Να σας χαιρετήσω όλους με ιδιαίτερη συμπάθεια. Και δεν θέλω να πω η παλιά μου φίλη, αλλά η φίλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, που με κάλεσε με τιμά ιδιαίτερα. Ήρθα λοιπόν εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού για να μιλήσω για το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Σπιτικού Ιστορίας. Εγώ παίρνω το λόγο ως πρόεδρος της Επιτροπής Επαφής ε, που το Προεδρείο του Κοινοβουλίου όρισε για να μπορέσουμε να βρούμε τη σχετική υποστήριξη τους ε, και τους σπόνσορ ε, διαφόρων τομέων και εντός και εκτός κοινοβουλίου στον πολιτικό τομέα. Ούτως ώστε το σχέδιο να καταστεί εφικτό. Αν θέλετε να ακούσετε τα προηγούμενα, δηλαδή την ιστορία του σπιτιού της ιστορίας, θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ στο παρελθόν. Δηλαδή είχαμε πολλές εκλογές ε, που μεσολάβησαν από τη στιγμή της απόφασης και μετά. Και η ιστορία γινόταν σαν το, μύθο του, σαν το παραμύθι του γεφυριού της Άρτας. Δηλαδή δεν τελείωνε ποτέ αυτή η ιστορία. Ε, κάθε φορά που γινόταν, μεσολαβούσαν εκλογές ή οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, ο μετρητής ε, πήγαινε στο μηδέν. Και ο Χάνσγκερ Πέτερινγκ, που ήταν πρόεδρός μας ε, στο Κοινοβούλιο το 2007, στον πρώτο του λόγο έθεσε το σπίτι της ιστορίας ως προγραμματική πλέον διακήρυξη και για το κοινοβούλιο και για την εκλογή του. Μία ιδέα που μας γοήτευσε πολλούς, κυρίως όσους γνωρίζαμε το σημείο αναφοράς, το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας, που τότε ήταν στη Βόνη το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας που είχε λάβει και το βραβείο του καλυτέρου μουσείου της Ευρώπης. Ένα βραβείο που όταν η Ντόρι Σπακ και εγώ εδρεύαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και εγώ ήμουνα πρόεδρος της, κοινο... της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, τέλος πάντων τότε του είχε δοθεί ένα βραβείο σε αυτό το μουσείο. Ένα αξιοθαύμαστο μουσείο το οποίο το επισκεπτόμασταν πολύ συχνά γιατί τότε πηγαίναμε συχνά στην Βόνη και ελπίζω και πολλοί ε, κόσμος να συνεχίζει να το επισκέπτεται και έχει μάλιστα σήμερα και ένα παράρτημα στη Λιψία. Αυτό ήταν το σημείο αναφοράς ε, που είχαμε ε, κατά νου και θεωρούσαμε ότι προσπάθειες παρόμοιες για αυτό το σπίτι της ιστορίας, δηλαδή τι ήταν αυτό το, αυτό το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας, ήταν και το σπίτι υποθήκης κληρονομιάς ε, της ε, γερμανικής ιστορίας. Και εμείς ε, και στην Ολλανδία προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και εκεί να βάγει σαν η ιστορία. Πρέπει να πω ότι το, σχέδιο το εξετάζαμε με πολλές απορίες, πολλά ερωτηματικά. Ξέραμε ότι ήταν κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρήσαμε λοιπόν, ακριβώς επειδή ήταν ένα δύσκολο σχέδιο, ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε τότε ήταν, μα είναι δουλειά του κοινοβουλίου, ε, ένα κοινοβούλιο μπορεί να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία ή είναι άλλες οντότητες που θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα. Ρωτώ λοιπόν εγώ. Εγώ τώρα σας είπα, διακόπτει την πρότασή του ο κύριος Μαρτίνης και αρχίζει μια καινούρια, ότι εδώ και 15 χρόνια είναι στα σκαριά αυτό το μουσείο και εδώ και 15 χρόνια δεν κατάφερε να γίνει τίποτε. 20 χρόνια συζητιέται το θέμα της Ευρωπαϊκής, του Μουσείου Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Βρυξέλλες και 20 χρόνια που δεν, ε, που δεν πετυχαίνει αυτό το σχέδιο. Αφενός γιατί είναι μπερδεμένο και δεύτερο χρειάζεται να μαζευτούν όλοι οι ιστορικοί από όλη την Ευρώπη, όλοι οι διευθυντές από όλα τα μουσεία της Ευρώπης. Ε, μα αυτός ο τρόπος είναι ένας από τους πολλούς ε, για να ε, δολοφονηθεί το σχέδιο στα γενοφάσκια του. Και τώρα το κοινοβούλιο, με, όχι φυσικά όχι το κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα και φυσικά άμα είναι δουλειά του Συμβουλίου να φτιάξει το μουσείο, το, το σχέδιο να βάγει, είναι σίγουρο. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να έχουμε 27 χώρες που θα πρέπει να συμφωνήσουν να φτιάξουν ένα μουσείο όπου ο καθένας επιμένει να διηγούνται τη δική του ιστορία. Αυτά για, για τις προηγούμενες αποτυχίες. Αυτό το οποίο θέλουμε λοιπόν σήμερα είναι το Προεδρείο να αποφασίζει ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτό το σχέδιο και όσο θα προχωράει αυτό το σχέδιο τότε θα εμπλέκονται άλλα θεσμικά όργανα, πιο συγκεκριμένα η Κομισιόν, το Συμβούλιο, όταν έρθει η ώρα και οι βελγικές αρχές οι οποίες είτε είναι ε, δημοτικές, ε, είτε περιφερειακές, ομοσπονδιακές, το βελγικό κράτος, ας πάνω. Αυτός είναι ο καρπός της προηγούμενης εμπειρίας και των αποτυχιών που είχαμε μέχρι τώρα. Εμείς λοιπόν συνειδητοποίησαμε απόλυτα ότι αν δεν έκανε το κοινοβούλιο αυτή τη δουλειά δεν θα την έκανε κανένας. Υποστηρίχθηκε λοιπόν από όλες τις πολιτικές ομάδες η πρόταση και το Προεδρείο αποφάσισε να ξεκινήσει την πρωτοβουλία τον Δεκέμβριο του 2007. Και τότε με διόρισαν, <laughs> μου ανέθεσαν ένα αξίωμα που εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τι ήτανε. Διευκολυντής ελληνικά θα ήτανε, «φασιλιτατέρ» στα γαλλικά. Και δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό λέει ο κύριος Μαρτίνες τι ήτανε. Και περάσαμε λοιπόν σιγά σιγά σκοπέλους, προβλήματα, σκεπτικισμούς, δισταγμούς και καταφέραμε αρκετά πράγματα. Λοιπόν το πρώτο ήτανε ο πρώτος μας στόχος ήταν να συλλάβουμε γενικό το σχέδιο, να δημιουργήσουμε μία ιδέα. Επιλέξαμε λοιπόν εννέα, εννέα ιστορικούς πολύ γνωστούς, έγκυρους ιστορικούς και με διαφορετικές θέσεις. Από τον Διευθυντή των Μουσείων του Βατικανού μέχρι τον ε, Διευθυντή των ε, Μουσείων ε, της Μασονίας. Κόσμος λοιπόν με μεγάλη εμπειρία για το τι εστί η ιστορία και το τι είναι τα διάφορα μουσεία, τα πιο κλασικά, τα πιο μοντέρνα κλπ. Και εγώ λοιπόν συμμετείχα σε αυτήν την ομάδα εργασίας εκπροσωπώντας το κοινοβούλιο. Ήταν μία εμπειρία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί πρώτα απ' όλα εγώ ποτέ μου δεν συμμετείχα σε μία ομάδα διανομένων αυτών των, ε, αυτού του μεγέθους. Και η δουλειά μου ήταν κάθε φορά να τους προσγειώνω και να τους λέω κοιτάστε δεν θα ξαναχτίσουμε το Λούβρο ή το British Museum ή το Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο. Πρέπει να κάνουμε κάτι το ταπεινό τέλο πάντων με μεγάλο περιεχόμενο. Και το πιο σημαντικό ήταν να καταλάβει κανείς ότι αυτό το οποίο θα έβγαινε από αυτήν την συνεδρίαση από αυτή, δεν θα ήτανε οι νόμοι του Μουησί. δεν θα ήταν οι πλάκες του νόμου. Απλώς έπρεπε μια πλατφόρμα να βγει, ένα πλαίσιο. Και το σπίτι γερμανικής ιστορίας που είχαμε κατά νου, ε, μας οδηγούσε να φανταστούμε ένα μουσείο το οποίο θα λειτουργούσε ως μουσείο της ιστορίας Ευρώπης από το 1945 και μετά. Δηλαδή η ιστορία που είχαμε μέχρι τότε, καταστροφής ε, πολέμου σφαγών, κατάφερε μέσα από ένα θαύμα της πολιτικής μεταξύ των άλλων να ξεπεράσει τον πόλεμο για την ειρήνη και να περάσει τη σύγκρουση για την υπέρ της ενσωμάτωσης. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος του Μωσίου. Πώς καταφέραμε δηλαδή να οικοδομήσουμε αυτή την Ευρώπη ειρήνης ειρήνης που καθόρισε τη σταθερότητα και η σταθερότητα ένα άνευ μια ανευπροηγουμένου κοινωνική πρόοδο. Αλλά βέβαια Οι συνεισφορές λοιπόν όλων αυτών των ιστορικών, μουσιολόγων, όλων αυτών των μεγάλων διανοουμένων οδήγησε στο να πούμε ότι ορίστε δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι το μουσείο ξεκίνησε το 45 χωρίς να ξέρουμε πώς φτάσαμε στο 45. Οπότε το πλαίσιο, κατά προσέγγιση βέβαια, έλεγε ότι το, τα τρία τέταρτα του, του μουσείου θα πρέπει να είναι αφιερωμένα στο ξεπέρασμα του πολέμου υπέρ της ειρήνης για να καταλήξουμε στο που είμαστε σήμερα. Και θα έπρεπε να έχουμε και ένα τέταρτο όπου θα λέγαμε τα ουσιαστικά της ιστορίας του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και ίσως ακόμη και ένα κομμάτι της ιστορίας του τέλους του 19ου και ίσως επίσης και καμία ελάχιστη αναφορά από την κλασική εποχή μέχρι σήμερα. 5% λοιπόν στην ιστορία μέχρι την σύγχρονη ιστορία, μέχρι τη μοντέρνα συγγνώμη ιστορία, ένα 15% για τον 20ο αιώνα. Και μετά η σύγχρονη ιστορία. Αυτό δηλαδή που ζούμε εδώ και 70 χρόνια. Το δεύτερο μισό λοιπόν του 20ου αιώνα και τον 21ο αιώνα. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι ένα μουσείο ιδιαίτερα interactive, διαδραστικό, και θα έπρεπε ένα μέγα μέρος να είναι περιοδεύουσες εκθέσεις. Να έχει σίγουρα μόνιμες εκθέσεις, αλλά κυρίως περιοδεύουσες εκθέσεις, διότι το μουσείο θα πρέπει, έχει δηλαδή την αποστολή να είναι συνδεδεμένο με εκατοντάδες ε, μουσεία, πολιτιστικούς ε, οργανισμούς, πανεπιστήμια, οπότε θα έπρεπε να ταξιδεύει για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί τι φτιάχνει. Επίσης, μια άλλη πτυχή του μουσείου είναι η πολυγλωσία. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι ένα μουσείο πολύγλωσσο σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Είναι οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης, όχι βασικά ομιλούμενες όπου οι συνεδριάσεις μας γίνονται σε δύο-τρία γλώσσες και μόνο, μόνο το κοινοβούλιο είναι πολύγλωσσο. Θα σας δώσουμε βέβαια και ένα χαρτί με ένα χρονοδιάγραμμα. Και όταν αποφασίστηκε η έγκριση όλης αυτής της ιδέας ως modus operandi, ορίστηκε ένα διοικητικό συμβούλιο, ακαδημαϊκό διοικητικό συμβούλιο το 2009. Και ως προς τους ε, σπόνσορες, πρόεδρος παραμένει ο κύριος Πέτερινγκ, εγώ είμαι αντιπρόεδρος, αλλά υπάρχουν και πολλές προσωπικότητες σε αυτό το συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργό ε, της ε, Περιφέρειας των Βρυξελών, η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και η κυρία Παλιαδέλη, ο κύριος Λαμασούρ, πρόεδρος Επιτροπής Προϋπολογισμών, η αρμόδια επίτροπος, δηλαδή η κυρία Βασιλείου. Συμμετέχει ο κύριος Χιούτε, που είναι ο διευθυντής του γερμανικού σπιτιού ιστορίες. Ο κύριος ε, ε, Μπόρτσικ, ο οποίος είναι ο αντιπρίτανης ε, του Πανεπιστημίου της ε, Βαρσοβίας και μετά έχουμε και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο που συμμετέχουν περίφημοι ιστορικοί και διευθυντές μουσείων. Αυτά μέχρι τον Φεβρουάριο που άρχισε να λειτουργεί, Φεβρουάριο 2009. Δημιουργήθηκε μετά η ομάδα επαφής. για να προασπίσουμε το σχέδιο μέσα στο Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα. Τον Ιούνιο το 2009 αποφασίστηκε το πού θα εδρεύει το μουσείο. Το μουσείο θα εδρεύει σε ένα κτίριο που αγόρασε το κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό με εξαιρετικέ συνθήκες από τις βελικικές αρχές και είναι ένα κτίριο 100 μέτρα να, πιο πίσω και δείχνει ο μιλητής. Είναι το κτίριο Eastman. Είναι ένα μοντερνιστικό κτίριο ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά, είναι ένα κτίριο το οποίο δεν μπορούμε να το πειράξουμε διότι είναι διατηρηταίο, αλλά όμως αυτό το κτίριο παλιότερα ήταν οδοντιατρική σχολή και πρέπει να ξαναφτιαχτεί εντελώς μέσα. Αποφασίστηκε λοιπόν το Προεδρείο να ξεκινά προκηρύξει έναν διαγωνισμό αρχιτεκτόνων για την ανάπλαση του κτηρίου. Και μας έδωσαν και είχαμε απίθανες απαντήσεις. 130 αρχιτεκτονικά γραφεία, αρχιτέκτονες που απάντησαν Και όταν τους εξηγούμε περί τίνος πρόκειται, μείναν 26. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν πολυεθνικό χαρακτήρα. Είναι 4-5 χώρες που συνεργάζονται και έχουν ήδη σχέδια φιλόδοξα στον ίδιο τομέα. Προχωρήσαμε και από τους 26 προεπιλέξαμε 12 που έχουν τώρα την ε, ευθύνη πλέον να δουλέψουν αντεπροέκτο, δηλαδή με σχέδια πλέον. Μουσιόλογοι λοιπόν συνεργάζονται και σε αυτά τα σχέδια και θεωρήσουν μετά από αυτά τα σχέδια που θα μας δώσουν ποια είναι τα δύο-τρία σχέδια που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και το Προεδρείο θα συζητήσει με τους μεν και με τους δε μεταξύ των άλλων για να δούμε και τι θα στοιχίζει δηλαδή. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Ο προϋπολογισμός είναι ένα θέμα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ξέρουμε ότι οι βελγικές αρχές θα συμμετέχουν σημαντικά, ήδη δεσμεύτηκαν με διάφορα εκατομμύρια, αλλά δεν είναι σαφές τι θα κάνει το κοινοβούλιο. 1,5 εκατομμύριο έχει φέτος. Αυτό χρειάζεται για το σχέδιο, τα προσχέδια κλπ και το 2011 θα προχωρήσει σημαντικά, ελπίζουμε. Στις 23 αυτού του μήνα έκλεισε η προθεσμία σχετικά με το προσωπικό που θα ασχολείται ένας διευθυντής με πιο μόνιμο χαρακτήρα και οκτώ επιστήμονες που θα έχουν ως αρμοδιότητα να ε, συνοδεύουν τους συνεργάτες κλπ. Με συμβόλαια τριών ετών. διότι μέχρι στιγμής όλα αυτά λειτουργούν με προσωπικό του Κοινοβουλίου, το οποίο μερικώς ε, χρήσιμο, ασχολείται με αυτό το σχέδιο, το οποίο θα πάρει πολύ καιρό. Και πραγματικά παίρνει χρόνο όλη αυτή η ιστορία. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν. 4.000 τετραγωνικά μέτρα το που θα έχει το μουσείο για τις μόνιμες εκθέσεις, 800 για τις εποχιακές εκθέσεις και 200 για τα γραφεία, τη ρεσεψιόν κλπ. Οι αποθήκες ε, δεν θα είναι φαντάζομαι στο κτίριο αλλά στο κοινοβούλιο το ίδιο όπου υπάρχουν άπειρα υπόγεια και μπορούμε να αποθηκεύσουμε οτιδήποτε. Εμείς ε, τελειώσαμε τώρα με τις υποψηφιότητες και το Προεδρείο θα αποφασίσει ποιους υποψήφιους θα επιλέξει. και έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι η ομάδα θα πρέπει να είναι και επιστημονικά ισορροπημένη και εθνικά ισορροπημένη και τα φύλλα θα πρέπει να είναι ισορροπημένα η εκπροσώπησή τους. Και να μην ξεχνάμε και τον προϋπολογισμό. Διότι Ήδη κάποιοι συνάδελφοι από την ομάδα μου έχουν αρχίσει και μουρμουρίζουν και λένε ότι ορίστε υπάρχουν τόσα λεφτά που είναι αστείο ποσό δηλαδή. 2,5 εκατομμύρια. Αλλά αυτά τα 2,5 εκατομμύρια όταν δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο τελικός προϋπολογισμός του σχεδίου δεν ξέρουμε σε πόσο θα τα χρησιμοποιήσουμε. και έχουμε και ένα σωρό επιστήμονες οι οποίοι μελετούν, επιστήμονες δηλαδή, αν η δομή του κτηρίου αντέχει να ρίξουμε έναν ή δυο ορόφους από πάνω και άμα δεν αντέχει λοιπόν η δυο απο πανω και αμα δεν αντεχει λοιπον η δομη του, σπιτιού άλλους δυο ορόφους ε, τότε πρέπει να ξοδέψουμε ακόμη παραπάνω. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τα 30 εκατομμύρια φυσικά όλα αυτά στο χρόνο, τα 3-4 χρόνια. Διότι ξέχασα να σας πω ότι θέλουμε να εγκαινιαστεί το μουσείο το 2014 που θα έχουμε έναν αιώνα δηλαδή από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Θέλουμε λοιπόν ένα μεγάλο σπίτι, ένα μουσείο που θα το επισκέπτονται όλοι όσοι έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που θα λειτουργεί και συμπληρωματικά με το κέντρο επισκεπτών που ασχολείται μόνο με τους επισκέπτες του Κοινοβουλίου και θα το επισκέπτονται και εκατοντάδες χιλιάδες τουριστών που έρχονται στις Βρυξέλλες. Και πριν από κανένα μήνα εγώ διάβασα μια ολόκληρη σελίδα στη Μόντα όπου έγραφαν ότι είναι σκάνδαλο να μην έχουμε ένα μουσείο για την Ευρώπη. Ποιο ξέρει, ίσω τα, τα, μάθανε από, από Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε τις αποτυχίες των προηγουμένων προσπαθειών όπου μπλέχτηκαν οι οικογένειες των ε, μεγάλων βέλγων πολιτικών του καιρού εκείνου, η βελγική κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων. ξεπεράστηκαν οι στιγμές του παραλογισμού και πρέπει να προσγειωθούμε και να αρχίσουμε να συζητούμε τι συλλογές θα βάλουμε εκεί μέσα. Και η Επιτροπή του Μουσείου θα πρέπει να αποφασίσει. Διότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει στο τι βάζουμε και τι δεν βάζουμε στο μουσείο ή αλλιώ ξαναπάμε πάλι στο μηδέν. Όπως ε, όταν παίζουμε στον Κρινιάρι που γυρνάμε πίσω. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε Πώς θα φτιάχνουμε όλα αυτά. Ποια θα είναι η παραμουσιακή δραστηριότητα που θα οργανώσουμε ερευνήτες, πανεπιστημιακούς που μπορούν να έρθουν και να κάνουν, και να κάνουν μια διατριβή, τι τεκμηρίωση θα πρέπει να τους διαθέτουμε και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις νέες τεχνολογίες τις πιο απίθανες για να έχουμε πραγματικά καλά αποτελέσματα. Τελειώνω λέγοντας ότι είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, είναι και ιδιαίτερα γοητευτικό θα έλεγα, θελκτικό σχέδιο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μη επιστροφής. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως εγώ από αυτή την Επιτροπή και γνωρίζοντας και την κυρία Πακ και την άλλη με συνάδελφο από την Επιτροπή των Σπονσόρων, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει η Επιτροπή σας να δεσμευτεί έντονα και να συμμετέχει. Ίσως και ως Επιτροπή και θα έπρεπε να γίνονται και συνεδριάσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο όπου να μπορούμε να συζητάμε, να μαζεύουμε ιδέες. Αλλά όταν αυτό ανοίξει, Όταν ξεκινήσει μόνο κάτι τέτοιο θα πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα γιατί άμα αρχίσει όταν ήδη θα έχει προχωρήσει το μουσείο θα είναι πολύ αργά. Βέβαια κυρία Πάκ, εσείς έχετε τώρα άλλες πολύ σημαντικές αρμοδιότητες, ελπίζω να μην χάσετε το πάθος σας για αυτή την πρωτοβουλία, ούτως ώστε αυτό το σχέδιο να ευωδώσει ευχαριστώ τον Τόρις Πάκ, ευχαριστώ και όλους τους υπόλοιπους για την υπομονή σας, ευχαριστώ Μιγγέλ. Ακούσατε όλες τις εξηγήσεις, θα λάβετε και ε, σχετικό έγγραφο. Το πρόγραμμα έχει φτάσει σε σημείο που δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πια πίσω. Αυτό είναι καλό, διότι έχουμε, ε, έχουμε αναμείνει πολύ και πιστεύουμε ότι έτσι κλείνουμε ένα σημαντικό κενό. Χρειαζόμαστε γνώση για τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια και λίγα μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία για το θέμα της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι το σπίτι Ευρωπαϊκής Ιστορίας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά, τουλάχιστον σε αυτούς που θα το επισκεφτούν. Και αν χρησιμοποιηθούν όλες οι νέες τεχνικές που υπάρχουν σήμερα, όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες για... που μπορούν να βοηθήσουν να κάνουν πιο καθαρά τα πράγματα αυτά στον επισκέπτη, Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά και έχεις δίκιο. Είναι η υποχρέωση του θεσμικού αυτού οργάνου να αναλάβει το θέμα και θα έπρεπε η Επιτροπή μας να ε, αγωνιστεί για το θέμα αυτό. Η συνάδελφος Παλιαδέλη και εγώ συμμετέχουμε ε, ώστε και η Κωνσταντζε Ίνσελ από τη γραμματεία μας ε, συμμετέχει ε, στις επαφές. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε πιο εντατικά με το θέμα αυτό όταν επιλεγεί αρχιτέκτονας. Τότε ως Επιτροπή θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τι μορφή θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο. Και μόλις είπα στον Σίμεν ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω του χρόνου να εκπονήσουμε έκθεση πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Έτσι θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά και θα φανεί η σχέση ε, του Μουσείου με την Επιτροπή μας. Ο κύριος Φίσας ζήτησε το λόγο, η κυρία Παλιαδέλη και Πέλα Παρακαλώ, κύριος Φίσας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Καταπληκτική πρωτοβουλία αυτό το Μουσείο της Ευρώπης. Πολλές φορές εμείς παραπονιόμαστε γι' αυτό την ε, έλλειψη εικόνας που έχει η Ευρώπη, αυτή τη δυσκολία που έχουμε να πουλήσουμε την παλιά μας Ευρώπη στους νέους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ καλό η Ευρώπη να κάνει κάτι το δυνατό και φανταχτερό όπως είναι αυτό το μουσείο. Τώρα κοιτάζω εγώ αυτό το έγγραφο που μόλις ε, ε, μας ε, μοιράσατε και ήθελα να ρωτήσω έκλεισε το μουσιακό σχέδιο διότι μπορεί να υπάρχουν και διάφορες ανισότητες στην ιστορία της Ευρώπη. Ξέρετε ότι την ιστορία συνήθως τη γράφουν οι νικητές ε, επί των νικημένων. Λοιπόν μπορεί να υπάρχουν ε, ανισότητες, όχι μόνο θεσμικού, ε, θρησκευτικού χαρακτήρα, συγγνώμη, μπορεί να υπάρξουν και εθνικισμοί βάριου τύπου και δύσκολο είναι πολλές φορές να καταλήγει κανείς σε μια κοινή αντίληψη. Πολλές φορές είναι στο και, μέχρι και αδύνατον. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους. Γιατί την αλήθεια ε, πρέπει κάπου να τη βάζουμε κι αυτήν. Άμα ξεπεράστηκαν αυτές οι δυσκολίες, εγώ θεωρώ ότι είναι μια καταπληκτική ιδέα και η Επιτροπή Πολιτισμού είναι έτοιμη να συνεργαστεί απόλυτα μαζί σας. Ευχαριστώ. Κυρία Παλιαδέλη. Ε, Ευχαριστώ κυρία. Χαίρομαι ιδιαίτερα ότι μου δόθηκε η μεγάλη ευκαιρία να μετέχω με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής ε, στο, συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σπίτι της Ιστορίας και ομολογώ ότι χάρη στην σημερινή παρουσίαση του κυρίου Μαρτίνες συνειδητοποίησα την πικρή ιστορία που κρύβεται πίσω του. Ότι 20 χρόνια προσπαθεί ε, προσπαθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το πραγματοποιήσουν. Χαίρομαι ακόμη λοιπόν περισσότερο ότι μετέχω σε μια φάση όπου τα πράγματα φαίνονται να είναι πιο θετικά. Ε, διάβασα με πολύ προσοχή τους βασικούς προσανατολισμούς ε, the conceptual basis για αυτό το μουσείο και ομολογώ ότι οι εννέα ιστορικοί που το συνέταξαν κάναν πολύ μεγάλη δουλειά. Εκτιμώ ωστόσο, και εδώ είναι περισσότερο ερώτηση παρά παρατήρηση, ε, ότι το, το, το, ιστορικό, το, το σενάριο καλύτερα της έκθεσης θα πρέπει να ξαναγραφεί, ε, κύριε Μαρτίνες, ε, με έναν τρόπο που θα βοηθήσει τους μουσιολόγους να, στήσουν, να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα που θα είναι η περιγραφή των αντικειμένων ε, που θα συμμετάσχουν, που θα εκτεθούν προκειμένου να υποστηρίξουν την ε, ε, έκθεση. Χαίρομαι ιδιαίτερα ότι το 1945 και μετά είναι πραγματικά ορόσημο για την Ευρώπη και την Ενωμένη Ευρώπη και νομίζω ότι με αυτήν την κατανομή κυρίως τον 20ο αιώνα τέλη του 19ου μέχρι και το, μέχρι τα μέσα του αιώνα είναι πολύ σωστή γιατί έτσι αποφεύγουμε ίσως τις ανησυχίες τις οποίες διατύπωσε προηγουμένως ο κύριος ε, Φίσας. Ε, ωστόσο εκτιμώ ότι το 5% ως παρελθόν είναι πραγματικά πολύ λίγο για το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν της Ευρώπης και εκτιμώ ότι ένα τέτοιο παρελθόν και σας έχω δώσει ένα σημείωμα ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι μόνο η ιστορία των ιδεών ε, προκειμένου να αντιπροσωπευθεί αυτό το 5% κοινό πολιτιστικό παρελθόν. Ε, είμαι μαζί σας, <laughs> θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να κάνουμε πραγματικότητα το 2004 αυτό το μουσείο. Να είστε καλά. Euh, Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση που μοιάζει με αυτή τη συναδέλφου. Δηλαδή, εφόσον είναι σημαντικό να υπάρχει μία ε, ιστορία για μετά το 45 η Ευρώπη υπήρχε και πριν το 45 και ελπίζω ότι θα καλύψουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διότι και ο Μεσαίωνας και η, ανα, η ε, αναγέννηση θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, σε αυτό το χώρο. Επίσης θα ήθελα να ξέρω αν ο Εντγκάρ Μωράν παραδείγματος χάρη πεπισμένος Ευρωπαίος έχει περιληφθεί και αν όχι ε, εάν πρόκειται να έρθετε σε επαφή μαζί τους, να σας πει και αυτό στη δικιά του γνώμη, η οποία σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσα. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν το θέμα της απεικιοκρατίας και της, ε, ε, του δουλεμπορίου θα ληφθεί επίσης υπόψη σε αυτό το ιστορικό παρελθόν της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριο Στόκης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ διότι το θέμα αυτό έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τον κύριο Μαρτίνες. Τον συγχαίρω θερμά, διότι η έκθεση αυτή μας δίνει μία πάρα πολύ καλή εικόνα ε, και ενημέρωση επί του προγράμματος αυτού. Εγώ είμαι Ανατολικοευρωπαίος, οπότε ε, θέλω να τονίσω μία συγκεκριμένη πτυχή, ε, διότι το έγγραφο που μας μοιράσατε, το έγγραφο αυτό, το κοίταξα στα γρήγορα, το ξεφίλησα και θα ήθελα να τονίσω ένα θέμα, δηλαδή η ιστορία της Ευρώπης, της ε, Μέσης και Ανατολικής Ευρώπης ε, πρέπει να παρακολουθεί ολοκληρωμένα διότι η Ευρώπη επί σειρά δεκαετιών έχει κατακαιρματιστεί και η ιστορική μας γνώση ε, υφίσταται ένα κατακαιρματισμό των γνώσεων. Για την Ανατολική Ευρώπη παραδείγματος χάρη έχουμε στην Ανατολική Ευρώπη παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει επίγνωση της ιστορίας της Δυτικής Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι δύο πτυχές να συγκεραστούν διότι διάβασα ότι αναφέρονται η ελληνική, η τουρκική, η ε, πολωνική μειονότηση μειονότητα αλλά προετών είχε υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της Ουγγαρίας εκ των οποίων ένα μέρος της χώρας απεκόπη υπήρξε μια ιστορική καταστροφή και στο έγγραφο αυτό δεν αναφέρεται η δικιά μας ιστορία θα πρέπει λοιπόν να τα συμπληρώσουμε αυτά η κυρία Ναβατήλοβα Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχέλ Άγχελ για την θαυμάσια παρουσία και για το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αφοσιωμένοι άνθρωποι στο πρόγραμμα αυτό. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε ε, να συμφωνήσετε ε, στο τι μας ενώνει και τι μας διαιρεί. Δηλαδή ποια είναι η κοινή μας ιστορία. Θα πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία κοινά και διαφορετικά για να τα περάσουμε σωστά στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ η κυρία Σάνεμπελ. Ευχαριστώ. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και πολύ σωστά ε, προχωρήσατε ε, και ευτυχώς που φτάσατε στο σημείο που φτάσατε παρόλες τις δυσκολίες. Νομίζω ότι ε, να επικεντρωθείτε για το μετά το 45 εξαρτάται από το σε τι θα αναφερθείτε για το παρελθόν. Ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα. Και μετά το 45 κοίταξα Ξεφίλησα το έγγραφο αυτό που αναφέρεται στα ουσιαστικά γεγονότα, αλλά τα ουσιαστικά γεγονότα είναι γνωστά στους ανθρώπους. Άρα αυτό που είναι σημαντικό είναι πώς θα το καταστήσετε ενδιαφέρον υπό την έννοια του μουσείου. Δεν είναι απλώς μια εξιστόρηση έγινε αυτό ή εκείνο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα θέμα. Και αυτό είναι η ευρωπαϊκή ενότητα, η συνένωση. Είμαι ε, σίγουροι ότι τα έχετε σκεφτεί αυτά, απλούστατα ίσως δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς το έγγραφο αυτό. Και αυτό είναι το θέμα όλων των εκθέσεων και ε, βεβαίως ε, το πρόβλημα ε, δεν είναι να βρείτε υλικό, θα έχετε πάρα πολύ υλικό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε και θα πρέπει να βρείτε ενδιαφέροντα παραδείγματα και εκθέματα κατά τρόπον ώστε να τονίσετε τα, τη διάφορη θεματολογία. θα ήθελα λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε για να ακολουθήσετε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ δημιουργικό για όλους, είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, έχουμε ακόμη έξι λεπτά για να απαντήσει ο εισηγητής. Νομίζω ότι δεν χρειάζομαι τόσο χρόνο, διότι ουσιαστικά ε, το θέμα είναι ε, ότι αναφέρεστε στο έγγραφο, αλλά μόλις δημοσιεύθηκε το έγγραφο αυτό, ιδίω στην ιστοσελίδα, υπήρξαν εκατοντάδες κριτικές αντιδράσεις, όλοι μας έλεγαν τι λείπει ε, και ε, ορισμένοι συνάδελφοι άλλωστε του Κοινοβουλίου, πολύ λίγοι, αλλά καθηγητές μας είπαν ότι ήταν σκανδαλώδες, ότι δεν είχαν περιλάβει αυτό ή εκείνο, οπότε γι' αυτό και επέμεινα και ο φίλος μου ο Φίσας θα αντελήφθη ότι αυτά τα οποία είπατε για τα ισπανικά θέματα δεν συμφωνούν με τη δικιά μου ιδέα διότι οι καθηγητές που το συζήτησαν ε, κάλυψαν ορισμένα θέματα και εγώ δεν έπρεπε να επέμβω προ προς το περιεχόμενο δεν ήταν αυτή ε, η εντολή μου δεν πρόκειται για την ιστορία του καθενός από εμά και των κρατών μας αλλά αυτό που είναι βασικό είναι να έχουμε ένα μόνιμο μουσείο και να τονίσουμε τις ε, άλλες εκθέσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να ε, εκφραστούν διαφορετικές απόψεις να υπάρξει μία θεματολογία για το παρελθόν, για, την, για το μεσαίωνα. Ξέρετε ότι πολλά από τα θέματα αυτά είναι ουσιαστικά για μας στην Ισπανία και θεματικά θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο των γυναικών, την ε, ε, κίνηση το, τη συνδικαλιστική, ε, τις ευθύνες των εργαζομένων. Εγώ δηλαδή αποδίδω μεγάλη σημασία στις μη μόνιμες εκθέσεις, οι οποίες θα είναι εκθέσεις που θα πάνε σε όλα τα μουσεία των χωρών μας όπου θα παρουσιάσουμε τα θέματα ε, και στις πιο μικρές χώρες. Και αυτό που είπε η κυρία Παλιαδέλη είναι πολύ βασικό. Δηλαδή ε, μία ανησυχία που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι δεν πρέπει να ανταγωνιστούμε με τα θέματα που καλύπτονται από μουσεία σε διάφορες χώρες όπου υπάρχουν πολύ ωραία μουσεία. Θέλουμε ένα μουσείο το οποίο θα δείχνει τι μας ενώνει χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε τα θέματα τα οποία μας χώρισαν. Είτε ήταν οικονομικά είτε ήταν θρησκευτικά θρησκευτικά ή ιδεολογικά, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο χώρο που θα αποδοθεί ε, ε, την, στον ε, πολιτισμό, είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως Πρέπει να υπάρξει χώρος ε, για την ε, αναγέννηση και για το Μεσαίωνα, αλλά αυτό θα είναι ένα πολύ ε, μικρό, ένας πολύ μικρός χώρος. Βεβαίως πρέπει να μιλήσουμε και για το μεσαίωνα και για την αναγέννηση αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας μία αίθουσα ε, για το μεσαίωνα και για την αναγέννηση είναι, ε, ε, είναι απαραίτητο. Αλλά στις 60 να υπάρχει μία και μία, διότι διαφορετικά οι Έλληνες και οι Ιταλοί μας φίλοι θα ήθελα να παρουσιάσουν όλοι ε, την αρχαιότητα. Αλλά μουσεία για την αρχαιότητα, όσο αιτιολογημένη και να είναι, υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη. Βεβαίως θα παραπέμπουμε στα μουσεία αυτά. Δεν μπορούμε να έχουμε σε ένα, ένα μουσείο για την ιστορία της Ευρώπης χωρίς ε, να τονίσουμε τι ε, αντιπροσώπευε η Ελλάδα και η οι ε, ε, ε, Λατίνοι διότι και η δικιά μου χώρα διότι και η χώρα μου η Ιταλία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να συμπεριληφθούν κατά τρόπον ώστε να μην δημιουργηθούν αντιδράσεις τώρα ο κύριος Τόκες, τον οποίον πολύ σέβομαι, μας έθεσε ένα πολύ βασικό θέμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να, να σκεφτούμε ένα τέτοιο μουσείο διαφορετικά. Δηλαδή γι' αυτό είπα ότι αν ξεκινήσουμε να μιλάμε το 1945 δεν μπορεί να μην μιλήσουμε για το Τριανό ε, για να ξέρουμε λοιπόν τι έγινε στο πρώτο ήμιση ε, του 20ου ε, αιώνα πρέπει να παραπέμψουμε στο τέλος του 19ου και στο πρόβλημα των μειονοτήτων που θα πρέπει να χαίρουν μια εξαίρετη θέση όπως θα πρέπει να περιληφθεί και το θέμα της μετανάστευσης. Δηλαδή εγώ όταν ε, βλέπω την ε, ε, γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα με ιταλικά, γαλλικά ονόματα, με ονόματα από το Μαγκρέμπ, αυτή είναι η Ευρώπη μας. Εάν δεν το καταλάβουμε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα είναι πάρα πολύ περίπλοκο έργο και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να πετύχουμε. Βέβαια η κυρία Χόνεγουελ πολύ σωστά μας τα λέει το πρόβλημα εδώ είναι πώς θα επιλέξουμε και τι θα επιλέξουμε. Αν είχαμε ένα μουσείο 50.000 τετραγωνικών θα τα καταφέραμε πολύ καλύτερα από ότι με ένα μουσείο 4.000 τετραγωνικών. Αν νομίζω ότι υπάρχει αρκετή καλή θέληση και πιστεύω ότι το μουσείο καλύτερο, πιο εύκολο θα ήταν για 12 χώρες από 27, αλλά δεν θα ήταν τόσο αντιπροσωπευτικό. Οπότε η πρόκληση αυτή μας δίνει την δυνατότητα να λάβουμε υπόψη και το, την Ανατολική Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να παρίσταται προμίας 20 ετίας. Οπότε και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Θα ήθελα έχετε πάρει το έγγραφο αυτό, διότι είναι σύντομο, αλλά νομίζω ότι με αυτό προσπάθησα να πείσω τους φίλους στην Επιτροπή Προπολογισμού ότι τους ζητούμε 2,5 εκατομμύρια για το 2011 και είναι λιγότερο από ό,τι ξοδεύουν για, για νερό, μεταλλικό νερό στις συνεδριάσεις μας. Ευχαριστώ. Βλέπετε ήταν πολύ ενδιαφέρον. Έχετε πολλούς φίλους εδώ και ε, όλοι οι συνεργάτες θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι 2 ε, και 2 Ιουνίου. Ευχαριστώ.